So, an. So, dear colleagues, welcome after the summer break for our... Καλώς ήρθατε για την πρώτη δημόσια ακρόαση για το ΦΠΑ σήμερα το απόγευμα. Τέσσερις ομιλητές ήρθαν εδώ στις Βρυξέλλες. Τους καλωσορίζω θερμά από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ο κύριος Γεώργιος Καρακατσάνης ο οποίος είναι επικεφαλής ε, του μέλους Νέιβεν Μάτες, του ιδιαίτερου γραφείου του, εκπρόσωπος ε, της PMP, e ο κύριος Γκέρχαρτ Χιούμερ, ο κύριος ε, Μάρτιν Γιάννετσεκ, εκπρόσωπος των τσεχικών αρχών, φορολογικών αρχών, και από την ε, Ένωση, η Γερμανική Ένωση ε, Ομοσπον... Αστυνομικών, ε, ο κύριος Σεμπάστιαν Φίτλερ. Δεν ε, ήρθε κανείς... Α, δεν ήρθε κανείς ακόμη. Α, ο κύριος Πόλιν δεν ήρθε. Άλλο μέλος ήρθε από την Κομισιόν όμως. Ωραία θα, θα παρέμβετε μετά τους τέσσερις προσκεκλημένους ομιλητές. Με μεγάλη χαρά θα σας ακούσουμε να παρουσιάζετε την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα, που είναι ε, προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και καταπολέμηση των απατών ΦΠΑ. Μέχρι 10 λεπτά θα έχουν χρόνο οι ομιλητές ε, νομίζω ότι θα ήταν πέντε αλλά είναι τέσσερις. Δέκα λεπτά λοιπόν θα κάνουν τις πρώτες παρατηρήσεις. Μετά θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής. Τα μέλη θα έχουν μέχρι τρία λεπτά χρόνο για την ε, ερώτηση και πέντε λεπτά θα έχουν μετά πάλι οι ομιλητές για να απαντήσουν και να κλείσουν. Ε, πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή της έκθεσης πρωτοβουλίας, τον κύριο Βάντερ Λάγεν, για να κάνει τις πρώτες παρατηρήσεις, προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω θερμά και εγώ και τους συναδέλφους και τους ε, ε, ε, ειδικούς εμπειρογνώμονες ως βάση Έχουμε την έκθεση, η ανακοίνωση της Κομισιόν από 7 Τετάρτου 16 για ένα πρόγραμμα δράσης στον τομέα του ΦΠΑ. Το σχέδιο έκθεσης από τη δική μου την πλευρά που διαβουλευτήκαμε είναι από 27 Τετάρτου. το Σεπτέμβριο θέλαμε να κλείσουμε το θέμα μετά από τις διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο, αλλά αναβλήθηκαν για το Δεκέμβριο. Βρήκαμε χρόνο λοιπόν να διοργανώσουμε και μία ακρόαση. Και με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων. Γνωρίζετε όλοι ότι το σύστημα ΦΠΑ με την έκτη οδηγία ΦΠΑ του 1993 χαρακτηρίστηκε μεταβατικό σύστημα και υπάρχουν πολλά προβλήματα γραφειοκρατικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προβλήματα απάτης στο εμπόριο ε, και στο διασυνοριακό επίσης και γι' αυτό οι προτάσεις έχουν ε, συζητηθεί με τα υπέρ και τα κατά. Τα φορολογικά θέματα όμως ε, θα πρέπει να αποφασίζονται με ομοφωνία. Υπάρχει μια πρωτοβουλία της τσεχικής κυβέρνησης από κοινού με την Ολλανδική Προεδρία να προτείνουν ένα νέο σύστημα της αντίστροφης επιβάρυνσης, της αντιστροφής της επιβάρυνσης, να δοκιμαστεί αυτό και επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, σε συνεννόηση με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή για θέματα ΦΠΑ συμφωνήθηκε να, να δοκιμαστεί ο, το ελεγκτικό συνέδριο εξέτασε το ΦΠΑ και θα πρέπει να δούμε ε, ποια είναι τα πιο κατεπήγοντα νομοθετικά προγράμματα και πώς ε, θα οργανωθεί καλύτερα η καταπολέμηση των απατών αυτών μαζί αν προσθεθούν και οι πληροφορίες που λείπουν σήμερα. Η αξιολόγηση της πρότασης One Stop Shop πώς κρίνεται από την, πώς, ποια είναι από τις ΜΜΕ και αν οι ΜΜΕ θεωρούν ότι θα είναι αποτελεσματικότερο το σύστημα reverse charge, αντισοφή δηλαδή της επιβάρυνσης για να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία. Τώρα προς την τσεχική φορολογική υπηρεσία σε φορείες, ε, εδώ θα ήθελα ο κύριος Γιάννετσεκ να μας μιλήσει για το μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης και την προθυμία της Τσεχίας και αν υπάρχει προετοιμασία για ένα τέτοιο πρόγραμμα και ερώτηση στον κύριο Φίντλερ από την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Εδώ μας ενδιαφέρει κυρίως το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις απάτες ε, στον ΦΠΑ. Και πώς κύριε Φίντλερ βλέπετε ε, να διαμορφώνονται οι δυνατότητες για μια ανταλλαγή διεθνών δεδομένων. Αυτά είναι κάποια θέματα. Δεν είναι όλες οι ερωτήσεις. Ε, ε, γενικά, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον αυτά, να ακούσουμε αυτά που θα μας πείτε. Και ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους και τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ τον Βέρνερ Λάγεν και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Καρακατσάνη για 10 λεπτά για να μας κάνει την παρουσίαση. Οι, οι, θα μιλήσουν μετά. Α, διαδικαστικά. Κύριε Πρόεδρε, κατάλαβα ότι θα, κάνετε, θα κάνει κάθε ομιλητής 10 λεπτά πρώτες παρατηρήσεις, μετά 3 λεπτά θα έχουν για τις ερωτήσεις και μετά οι ειδικοί θα μιλήσουν, θα απαντήσουν για 5 λεπτά. Προ, ε, προτείνω η εισαγωγική παρουσίαση να είναι μικρότερη για να έχουμε πιο πολύ χρόνο για τις απαντήσεις. Γιατί πέντε λεπτά για να απαντήσουν σε ένα σωρό ερωτήσεις που θα, έχει τεθεί στον, θα έχουν τεθεί στον καθένα είναι ε, ε, λίγο. Ενώ τα δέκα λεπτά ενδεχομένως να είναι πολύ. Πέντε λεπτά εισαγωγή προτείνω εγώ. Τρία λεπτά ε, ο κάθε βουλευτής και δέκα λεπτά να έχει μετά ο κάθε ε, εμπειρογνώμων για να απαντήσει. Τι λέτε, συμφωνείτε, τι λέει ο κύριος Λάνεν. Βεβαίως, θεμητό το αίτημα του συναδέλφου, αλλά έχουν προετοιμάσει τις ομιλίες τους οι εμπειρογνώμονές μας. Μπορούμε στο τέλος να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Μην ε, τους ζητήσουμε να είναι συντομότεροι στην αρχή. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί εμεί θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις τους, όχι να απαντάνε μόνο στις ερωτήσεις μας και ενδεχομένως να επιβεβαιώνουν αυτά που πιστεύουμε. Ο κύριος Λούκερ πάλι. Ναι, ε, εγώ κατάλαβα ότι είπατε ότι ήταν, ότι ήταν προετοιμασμένοι για πέντε λεπτά και μετά είπατε ότι ε, περιμένατε άλλον έναν ομιλητή. Όχι, δέκα λεπτά. Εγώ είδα ότι ήταν σημειωμένα 10 λεπτά και αυτό νομίζω είχαν ε, προγραμματίσει και οι ομιλητές μας. Οπότε καλύτερα είναι να ε, δώσουμε χρόνο περισσότερο στο τέλο. Στο τέλος. και αφού μιλήσουν και οι σκιώδεις, επειδή βλέπω ότι όπως και στην Ολομέλεια δεν είναι πάρα πολύ ε, ορισμένες φορές οι συνάδελφοι, Νομίζω ότι και σε διαδικασία catch the δεν θα φάμε πάρα πολύ χρόνο. Οπότε θα τα προλάβουμε όλα. Ο κύριος Καρακατσάνης πρώτος, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι επικεφαλής του γραφείου του κύριου Νεβερμάτες, μέλους του ε, Ελεκτικού Συνεδρίου. Ήταν υπεύθυνο τη έκθεση 24 του 2015 για την απάτηση στον τομέα του ΦΠΑ περισσότερη, χρειάζεται περισσότερη δράση. Να σας υπενθυμίσω ότι η έκθεση έχει ήδη παρουσιαστεί στο, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Κοινοβουλίου και στο Συμβούλιο στην αντίστοιχη ομάδα εργασία για τη φορολογία τον Απρίλιο. Κάναμε κάποιες συστάσει συστάσεις, οποίε από τις οποίες έλαβε υπόψη την υπόψη της Οικομισιόν, στο πρόγραμμα δράση τη ε, και στι προτάσει τη για την μεταρρύθμιση του ΦΠΑ. Για την αντιστροφή τη επιβάρηση μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσει σα καθώ και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα θεωρείτε. Το θέμα τη αντιστροφή τη επιβάρηση, ε, αν θέσει παραγράφου 88 και 89 τη ειδική έκθεση. Σα πω ποια είναι τα προβλήματα, ε, ποια είναι τα πορίσματά μα και ποιε είναι οι συστάσει μα. Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993 ήταν καλή για πολλού λόγου, αλλά δημιούργησε σημαντικές προκλήσεις στην συλλογή του ΦΠΑ, στην ίσπραξή του. Παλιότερα τα σύνορα εξασφάλιζαν ότι οι εισαγωγείς μπορούσαν να πάρουν τα εμπορεύματά του μόνο αφού είχαν πληρώσει το ΦΠΑ, ενώ οι εξαγωγείς επιτρεπόντουσαν να, επιστρα... να λάβουν επιστροφή ΦΠΑ, ε, μάλλον εξαίρεση ΦΠΑ, μόνο αν ε, τα τελωνία δεχόντουσαν τη διασαφή του. Μετά το 1993 οι έλεγχοι στα σύνορα αντικαταστάθηκαν από υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών ε, σε περιπτώσεις διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών. Οι εμπορευόμενοι πρέπει να υποβάλουν στις φορολογικές τους αρχές εκθέσεις ε, στις οποίες εντοπίζουν ε, τους αντιβαλλόμενούς τους στα άλλα κράτη-μέλη μέσω του αριθμού φορολογικού μητρώου τους. Οι ε, φορολογικές ε, αρχές του εξάγοντος κράτους μέλους ανταλλάσσουν αυτές τις, αυτά τα στοιχεία μέσω του συστήματος βίες και μάλιστα έχουν και λόγο να διαπιστώνουν την ειλικρίνεια των δηλώσεων αυτών γιατί αλλιώς θα χάνουν έσοδα. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός περιλαμβάνει και διοικητική συνεργασία ε, μεταξύ των, της, ε, στην οποία περιλαμβάνεται και η δημιουργία του Eurofisk. Ε, επίσης εισήγαγε και άλλα εργαλεία. Ζητώ συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη σας διακόπτω. Μιλάτε εξαιρετικά γρήγορα. Μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι δυνατόν. και άλλα, εργασία, άλλα εργαλεία διοικητικής συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών ε, με κατόπιν αιτήματος ή και όχι συν την δυνατότητα ταυτόχρονων ελέγχων σε δυο ή περισσότερα κράτη-μέλη με την παρουσία ε, ε, των φορολογικών αρχών από άλλα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα είναι ότι για αγαθά τα οποία εισάγονται από χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ονομάζεται Διαδικασία 42, μέσω ενό κράτου μέλου αλλά με τελικό προορισμό άλλο κράτο μέλο, οι ε, τελωνιακέ αρχέ δεν εισπράττουν πλέον ΦΠΑ. Σε αυτέ τι περιπτώσει, ο, ο, ο, το άτομο το οποίο ε, είναι ο τελικός προορισμό πρέπει να υποβάλει δήλωση ε, και ο, ο φορολογικός εκπρόσωπος του εισαγωγέα υποχρεώνεται να εισάγει στοιχεία επίσης στο σύστημα για τα εισαγόμενα είδη τα οποία στέλνονται στο άλλο κράτος μέλος μέσω του, του συστήματος βίας. Ε, όλο αυτό το σύστημα δημιουργεί προκλήσεις και προβλήματα στην ε, εισπράξη του ΦΠΑ και δημιουργεί παραθυράκια για απάτη. Αυτό που είδαμε στο πρόγραμμα δράσης της Κομισιόν για το ΦΠΑ είναι η ιδέα για μια ε, ενιαία ε, περιοχή ΦΠΑ, μια περιοχή ενιαίο ΦΠΑ ε, και ένα ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ το, τα οποία μπορούν να λύσουν ή να διευκολύνουν τη λύση των προβλημάτων. Η, ο έλεγχος μας ε, ανακάλυψε ότι συνολικά υπάρχει σύστημα για την καταπολέμηση της απάτης σχετικά με το ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τις διακοινωτικές συναλλαγές. Αυτό το σύστημα είναι πλήρε, πλήρες, αλλά έχει σημαντικές αδυναμίες που σχετίζονται πιο πολύ με την εφαρμογή του. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι σε μια ε, έρευνα, ένα ερωτηματολόγιο που στείλαμε σε όλα τα κράτη-μέλη, στις φορολογικές αρχές τους, για το κατά πόσο είναι αποτελεσματικές οι ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας που υπάρχουν, ε, οι περισσότερες αρχές εξέραν την ικανοποίησή τους για το πώς έχει στηθεί το σύστημα. Συμπλήν όμως, κατά τη διάρκεια της έρευνα, ε, εντοπίσαμε σημαντικές αδυναμίες στα έξι τουλάχιστον κράτη-μέλη τα οποία εξετάσαμε. Να σα πω ποιε είναι αυτές. Πρώτον, υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες σε ό,τι αφορά τις ε, διασταυρώσεις ε, μεταξύ τελωνίων και φορολογικών στοιχείων. Οι φορολογικέ αρχέ των κρατών μελών δεν έχουν ε, κίνητρα για να διαπιστώνουν και να διασταυρώνουν το κατά πόσον είναι αληθή τα στοιχεία που δηλώνονται από του εισαγωγεί. Δεύτερον, υπάρχουν προβλήματα ακρίβειας, ε, πληρότητας ε, και ε, εγκαιρότητας υπόβλησης των στοιχείων. Ε, επίσης, όταν εντοπίζονται ε, στις ανακεφαλαιωτικές δηλώσεις προβλήματα με αριθμούς φορολογικού μητρώου, ανύπαρκτους αριθμούς δηλαδή, πολύ συχνά τα κράτη-μέλη δεν κάνουν κάτι παραπάνω. Ε, επίσης, υπάρχουν αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες διαφόρων αρχών. Τέταρτον, η Eurofisk που είναι αποκεντρωμένη δομή ε, έχει μέλη ε, τα οποία όμως κάνουν ε, το καθένα τη δική του ανάλυση σε διαφορετικά κράτη-μέλη και με το δικό του software. Το αποτέλεσμα είναι ότι ανταλλάσσονται πάρα πολλά στοιχεία, μεγάλους όγκους στοιχείων, που όμως δεν έχουν σχέση με, ενδεχομένως με ε, απάτες. Πέμπτον, η Όλαφ και η Europol που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ε, δεν, έχουν ε, δεν έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών. Και τέλο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη δεν υφίσταται σύστημα συστηματική συλλογή και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων για, την, για περιπτώσει απάτη ΦΠΑ στι ενδοκινοτικέ συναλλαγέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έκθεσή μα. Γιατί πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο, αν είχαμε δηλαδή τέτοιου είδου πληροφορίε, θα διευκολυνόμασταν στο να ε, δημιουργήσουμε ε, μονάδες μέτρησης, ε, μέτρα για να μετρήσουμε την βελτίωση που επιτυχάνουμε. η... η, μια μελέτη έχει πρόσφατα ε, υπολογίσει στα 163 δισεκατομμύρια ευρώ τις απώλειες από μη σπραξή ΦΠΑ και ε, ε, παρόλα αυτά εντοπίζονται και εκεί ορισμένες αδυναμίες οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτό το νούμερο πάντως γενικά είναι πολύ μεγάλο το ποσό να πω η Κομισιόν κάνει προσπάθειες έκανε και μία μελέτη η οποία όμως δεν εκτιμά ε, παρκώς ε, την, το σύνολο της απάτης, το συνολικό ποσό απάτης. Μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες για αυτό το θέμα γιατί θεωρούμε ότι ε, δεν είναι, γιατί έχει αδυναμίες αυτή η μελέτη. Αυτό που μπορούμε να το μετρήσουμε μπορούμε να το βελτιώσουμε και χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία να μπορούμε να τα μετρήσουμε. κάποιες ε, διοικητικές αρχές, ιδιαίτερα στον Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο, ε, έκαναν σημαντική πρόοδο σε αυτό το τομέα και το αναφέρουμε στην, στο δική μας έκθεση με εφαρμοστικά μέτρα τα οποία βελτίωσαν πάρα πολύ την κατάσταση. Τώρα, ε, θα ήθελα να επαναλαβώ ότι το ελεκτικό συνέδριο έχει ω βασικό στόχο να εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνουμε γνώση λοιπόν ε, και σημειώνουμε το πρόγραμμα δράση τη Κομισιόν και όλε τι τελευταίε τη δράσει. Ε, ε, Ορισμένε από τι συστάσει που κάναμε τι έχει λάβει ήδη υπόψη η Κομισιόν. Παράγραφο 3-1 τη έκθεση συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά. Κάναμε διάφορε συστάσει, οποίε δεν θα επαναλάβω, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο αλλά η Κομισιόν δέχτηκε τις περισσότερες. Υπάρχει μία όμως την οποία δεν δέχτηκε. Παρόλο ότι την επαναλάβει δύο φορές ε, ε ο κ. Μάτες. Ζητήσαμε κάποιες νομοθετικές τροπολογίες που θα επέτρεπαν καλύτερες διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ φορολογικών αρχών και τελωνίων. Δεν είμαστε οι μόνοι που το ζητούν. Το γαλλικό ε, αντίστοιχο ελεκτικό συνέδριο ε, ζητά το ίδιο και μας ε, προβληματίζει το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν θέλει να αναλάβει δράση για αυτό το θέμα. Το ζητάμε εδώ και πολύ καιρό και εμείς και άλλα όργανα και άλλοι φορείς εκθέσει τους. Οι εμπειρογνώμες μάλιστα σε θέματα απάτης ΦΠΑ που συμμετείχαν στο, στην ομάδα φυσκάλης από το 2007 το είχαν συστήσει. Παρ' όλα αυτά χαιρόμαστε που η Κομισιόν σε δήλωσή της ε, αναφέρει ότι θα ξαναεξετάσει το θέμα αφού λάβει τις συστάσεις της ε, ομάδας του Project Fiscal 2020. Νομίζω ότι αυτές ήδη έχουν κατατεθεί. Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι το οποίο είπε ο κ. Μάτες ήδη θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε στενά την ε, πρόοδο και θα ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τακτικά όταν ε, μα ζητείτε. Εμεί μπορούμε να υποβάλουμε και γνωμοδότηση ή νομοθετικέ προτάσει, ε, αν μα ε, ζητηθεί, σε ό,τι αφορά τα θέματα καταβολή τη απάτη. Αυτή η γνωμοδότηση θα μπορούσε να καλύψει και θέματα τα οποία δεν έχουμε καλύψει τελευταίε μα εκθέσει. Για ε, παράδειγμα την αρχή του προορισμού στις ενδοκινοτικές ε, ε ανταλλαγές ε, και την αρχή του mini one stop shop. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή αυτή. Ο κύριος Γκέρχαρτ Χιούμερ έχει το λόγο τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Είμαι ευγνώμων που αποδίδεται μεγάλη σημασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό με καλέσατε εδώ. Ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα με τον ΦΠΑ. Ως έχει το σύστημα σήμερα. Όπως αναφέρθηκε, το σύστημα ΦΠΑ είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να μπουν σε, ε, στις επιχειρήσεις ΜΜΕ. Θα πρέπει να δούμε και ποιες, ποιοι είναι οι επαχθέστεροι κανονισμοί ε, όταν ε, ε, μεταξύ των πέντε επαχθέστερων ο ΦΠΑ συγκαταλέγεται πάντοτε στα ερωτηματολόγια. Χαιρόμαστε που μπήκε στην ημερήσια διάταξη το θέμα αυτό και θα προχωρήσει ένα πρόγραμμα δράσης για το ΦΠΑ, κυρίως σε ό,τι αφορά το θεματολόγιο απλούστευσης και η καταπολέμηση της απάτης, γιατί και η υπόθεση της απάτης είναι πολύ σημαντική. Γιατί οι φόροι που δεν πληρώνονται από τους απαταιώνες πληρώνονται από τους νομοταγείς ε, επιχειρηματίες. Ε, ε, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Τέσσερα θέματα θα θίξω. Το πρώτο είναι η απλοποίηση το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκλήθη να διευρύνει το mini one-stop shop και τις διαδικασίες παράδοση εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Είμαστε ευτυχείς διότι προτείνει την επέκταση η Κομισιόν για να συμπεριλάβει και όλες τις μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου. Αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζονται εύκολη πρόσβαση ε, στα συστήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Η ΜΜΕ δεν πρέπει να είναι εκείνες υπεύθυνε για την εφαρμογή του σωστού συντελεστή βάσει των πληροφοριών ενώ θα πληρώνουν πρόστιμα επειδή δεν τα έκαναν καλά. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι ΜΜΕ έχουν εύκολη πρόσβαση σε σωστές πληροφορίες. Δωρεάν επίσης πρέπει να μπορεί να βασίζεται σε αυτές τις πληροφορίες η μικρομεσαία επιχείρηση. Η Κομισιόν επίσης προτείνει ε, κάτω από ένα συγκεκριμένο κατόφλι ε, να μην χρειάζεται να ε, καταχωρίζονται σε άλλα κράτη-μέλη ή ΜΜΕ. Αυτό θα απλουστεύσει τις διαδικασίες των νεοφυών και μικρο, μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, δεν πρέπει να εξαιρούνται μόνο, να απαλλάσσονται μόνο οι νεοφυείς. Οι νεοφυείς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως άλλες μικρές επιχειρήσεις. Να μην γίνονται διακρίσεις μεταξύ νέων και υφισταμένων επιχειρήσεων. Το κατόφλι θα πρέπει να ισχύει σε όλες τις επιχειρήσεις κάτω από ένα συγκεκριμένο κύκλο εργασιών. Αλλιώς θα δημιουργηθούν εντάσεις και αθέμητος ανταγωνισμός. Επίσης είναι σημαντικό οι εταιρείε που ε, μπορούν να τύχουν απαλλαγών, να μπορούν, αν θέλουν, να εξαιρεθούν. Αν θέλουν δηλαδή να προχωρήσουν διαφορετικά, να μην είναι υποχρεωμένες να καταχωρίζονται ως μικρές επιχειρήσεις. Και βέβαια, συμφωνούμε με τις ιδέες της Κομισιόν σχετικά με τους ελέγχους στην χώρα προέλευσης και να ε, υπάρχει απαλλαγή για μικρές αποστολές από προμηθευτές τρίτων χωρών. Ένα άλλο θέμα είναι το ε, ενιαίο έντυπο ΦΠΑ. Πριν από δύο-τρία χρόνια είχε γίνει πρόταση από την Κομισιόν, αλλά δεν, ήταν, δεν ικανοποίησε τις ε, ΜΜΕ. Γιατί πάλι θα κατέληγαν σε διαφορετικά έντυπα ΦΠΑ, 28 συγκεκριμένα. Αν δεν υπάρχει εναρμόνιση, δηλαδή δεν έχει νόημα να αλλάξει το έντυπο αφού ε, θα αλλάξουν οι κανόνες, αλλά πάλι θα είναι διαφορετικά τα έντυπα. Τέλος, για την απλούστευση, συνεργαζόμεθα με την Κομισιόν για μια αναθεώρηση των ειδικών καθεστώτων για μικρές επιχειρήσεις ε, στα πλαίσια των ΜΜΕ, ε, απαλλαγές τα κατόφλια για την καταχώρηση, τη συμμόρφωση, μέτρα όπως λογιστική σε ταμιακή βάση και τα σχετικά καθεστώτα ε, ρυθμίζονται. Υπάρχουν διαφορές στην εφαρμογή στα κράτη-μέλη και υπάρχουν έτσι προβλήματα για τις ΜΜΕ. Ίσως θα πρέπει να το δουν πιο προσεκτικά αυτό. Εμείς δεν θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ε, ούτε η Κομισιόν έχει υποβάλει ακόμα συγκεκριμένες προτάσεις. Του χρόνου θα υποβάλει σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης. Τώρα, για την αντιστροφή της επιβάρυνσης και το σύστημα αυτό. Στο πρόγραμμα δράσης ε, αναφέρεται δύο φορές το σύστημα αυτό, αντιστροφής της επιβάρυνσης, πρώτα σε ένα προσωρινό σύστημα αντιστροφής επιβάρυνσης, που θα το εφαρμοστεί ως προσωρινό μέτρο για την καταπολέμηση της απάτης και δεύτερον ε, με, ως γενικευμένο σύστημα. Εμείς συμφωνούμε ότι μπορεί να συμβάλλει αυτό το σύστημα ε, στη, ε, στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ. Δεν είμαστε λοιπόν κατά του συστήματος αντιστροφής της επιβάρυνσης, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα συστήματα αντιστροφής της επιβάρυνσης εφαρμόζονται, εφαρμόζονται μόνο προσωρινά και μόνο από κάποια κράτη-μέλη θα δημιουργήσουν πρόσθετο κόστος και αβεβαιότητα για τις ΜΜΕ που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν διαφορετικούς πελάτες με διαφορετικούς τρόπους και αυτό συνεπάγεται και κόστος προσαρμογής και στην αρχή και στο τέλος. Γι' αυτό όλα μας τα μέλη είναι κατά ενός προσωρινού συστήματος αντιστροφής της επιβάρυνσης που θα εφαρμόζεται από κάποια κράτη-μέλη λόγω της νομιμικής ανασφάλειας, λόγω του αυξημένου κόστους και τον κίνδυνο για τις ΜΜΕ, αν γίνει λάθος. Αν δηλαδή ε, γίνει λάθος με τον αριθμό ΦΠΑ, ε, τότε το κόστος αυτών των συναλλαγών στο τέλος θα τα υπομιστούν οι ΜΜΕ και θα δημιουργηθούν νέα εμπόδια για την εσωτερική αγορά, αν εφαρμοστεί μόνο σε κάποια κράτη-μέλη. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει καινούργια παραθυράκια για φορολογικές απάτες, είτε μέσω άλλων χωρών ή χρησιμοποιώντας ε, με λανθασμένο τρόπο τον αριθμό ΦΠΑ. Και υπάρχει και ο κίνδυνος αυτά τα συστήματα να μπλοκαριστούν όταν πάμε σε οριστικό σύστημα. Εμείς είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και όλες οι εθνικές μας οργανώσεις λένε μην το κάνετε. Επόμενο, ε, οριστικό καθεστώς ΦΠΑ. Εμείς είμαστε υπέρ του οριστικού συστήματος ΦΠΑ που στηρίζεται στην αρχή της χώρας προορισμού, ε, όπως συμφώνησαν Κομισιόν και Συμβούλιο. Ε, θα πρέπει οι προμηθευτές από επιχείρηση σε επιχείρηση να φορολογούνται στα εμπορεύματα με τον ίδιο τρόπο όπως και οι εγχώροι. Το πιο σημαντικό για μας είναι η απλή πρόσβαση, η εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες ε, σε όλες τις χώρες. Τέλος, για τους φορολογικούς συντελεστές. Η Κομισιόν λέει ότι η μετάβαση προς την αρχή του προορισμού αφήνει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν το επίπεδο των συντελεστών. Εμείς δεν συμφωνούμε με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς αυτό, διότι η μεγαλύτερη διαφοροποίηση των συντελεστών ΦΠΑ θα στρεβλώσουν σοβαρά την ενιαία αγορά, ιδιαίτερα σε παραμεθόριες περιοχές, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και οποιαδήποτε συζήτηση για την αλλαγή των συντελεστών θα πρέπει να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο στην νέα αγορά, μη δημιουργώντας στρεβλώσεις ε, που τις είδαμε ήδη σε κάποιους τομείς εμπορευμάτων στο παρελθόν. Είμαστε λοιπόν θετικοί, θετικά διακείμενοι, αλλά ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην δημιουργήσουμε νέα προβλήματα για τις ΜΜΕ παρά τις καλές μας προθέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χιούμερ. Ο επόμενος ομιλητής, Γενικός Διευθυντής για τη Φορολογική Διοίκηση ο, την, ε, Τσεχία, ο κύριος Μάρτιν Γιάννετσεκ. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ για να συμμετάσχω στην συζήτηση όσον αφορά την απάτη σχετική με τον ΦΠΑ. Να σας παρουσιάσω ε, κάποια επιχειρήματα ε, τα οποία στηρίζουν το τσεχικό έτοιμο τόσο ώστε να εφαρμοστεί καθεστώς αντιστροφής επιβάρυνσης. Θα γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση η απάτη σχετική με τον ΦΠΑ γιατί ο ΦΠΑ είναι σημαντική πηγή εσόδων για τα κράτη-μέλη. Οπότε, ε, αν ε, συρρυκνώσουμε, αν μειώσουμε την απώλεια εσόδων, θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλούμε για 170 δις ευρώ κάθε χρόνο και κατά μέσο όρο ε, μιλούμε για το 15% του συνόλου της οφειλής για τον ΦΠΑ. Αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα, γιατί έτσι έχουμε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς και έχουμε επίσης πολλές περιπτώσεις ε, ε, της που της οποίας η μορφή ονομάζεται αλυσιδωτή απάτη. Αλλά επίσης έχουμε και ξεπλήμα χρήματος. Οπότε επίση υπάρχουν ε, στοιχεία το ότι το οργανωμένο έγκλημα επίσης εμπλέκεται. Δηλαδή, τα χρήματα που δεν αποδίδονται δεν χρησιμοποιούνται για καλό σκοπό. Αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους. Θα πρέπει επομένω ταχείως να βρεθεί κάποια λύση στο πρόβλημα. Έχουμε κάποια συμβατικά μέτρα τα οποία αποτελούν βραχυπρόθεσμη λύση. Αλλά δυστυχώς αυτά τα μέτρα δεν έχουν αποδώσει. Και ε, επίσης έχει αυξηθεί το διοικητικό άρθρος και για την διοίκηση αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχει υπάρξει η ιδέουσα ε, πρόληψη σαν αποτέλεσμα αυτών των μέτρων. Θα πρέπει επομένω να δούμε τι θα κάνουμε, τι μέτρα θα λάβουμε για να χτυπήσουμε το πρόβλημα στην ρίζα του. Θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο ένας των δύο συμβαλωμένων θα πρέπει να αποδίδει στις αρχές των ΦΠΑ. Και αυτός, σύμφωνα με το προτινόμενο σύστημα, θα είναι ο αποδέκτης των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών. Έχουμε εμπειρία σε σχέση με αυτό το σύστημα. Έχουμε ασχοληθεί με την καταπολέμηση της απάντησης και προσπαθούμε έτσι να χτυπήσουμε την αλυστοτή απάντηση στην ε, τσεχική δημοκρατία. Βέβαια έχουμε περιορισμένη επιτυχία. Γι' αυτό και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που να μην αντιβαίνει στην ιδέα, στη φιλοσοφία του ΦΠΑ. Πολλές φορές λένε ότι η αντιστροφή ε, της επιβάρυνσης υπονομεύει τον ίδιο το ΦΠΑ. Όχι, γιατί απλώς ένα στοιχείο μόνο ε, πειράζουμε με αυτό το σύστημα. Το υπόλοιπο σύστημα γίνεται πιο σταθερό και πιο ανθεκτικό Το υπήν. Επίσης υπάρχει φορολογική ουδετερότητα. Λειτουργούν διορθωτικοί μηχανισμοί όσον αφορά τον υπολογισμό του φόρου. Με τίποτα δεν έχουμε μόνο υπονόμευση του ΦΠΑ. Αντίθετα, γίνεται το σύστημα πιο στεγανό, πιο ασφαλές. Τι έχουμε κάνει στην Τσεχία. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την απάτη για τον ΦΠΑ και έτσι έχουμε θεσπίσει διάφορα μέτρα συμβατικού χαρακτήρα. Όμως δεν είχαμε καμία σημαντική επιτυχία στην καταπολέμηση της απάτης. Οπότε και τώρα θέλουμε να εφαρμόσουμε την αντιστροφή της επιβάρυνσης σε κάθε συναλλαγή που καλύπτεται από την οδηγία του ΦΠΑ. Και έτσι θεωρούμε ότι όπου έχουμε εφαρμόσει το σύστημα αυτό, έχει μειωθεί η ελιστοτή απάτη. Μπορείτε επομένω από τα στοιχεία που έχουμε να δείτε ότι το σύστημα αυτό αποδίδει, γιατί μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα περιορίσαμε σημαντικά την απάτη. Κατά 98% οπότε είπαμε για συγκεκριμένες αλλαγές θα μπορούσε να εφαρμόσει το σύστημα, αλλά αυτό δεν είναι η τέλεια λύση. Και αυτό γιατί τα σχετικά εμπορεύματα δεν κάνουν την εφαρμογή του μέτρου πάντοτε εύκολη. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κατόφλι υψηλό και για αυτό ζητούμε να εφαρμοστεί ένα πιλωτικό πρόγραμμα για ένα γενικευμένο σύστημα αντιστροφής της επιβάρυνσης. Μιλούμε για κατόφλι του ύψους των 10.000 ευρώ. Με ένα τέτοιο γενικευμένο σύστημα θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε για, από το πρόβλημα ανακλάδο της οικονομίας, κυρίως εκείνους που σοβεί η αλυσιδωτή απαραίτητη ο Λάγκεν το ανέφερε και μίλησε για το κατά πόσον είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Μπορούμε. Και επίσης μπορούμε να έχουμε επίσης την υποβολή εκθέσεων σε σχέση με ελεγχόμενες συναλλαγές. και ταυτοχρόνως έχουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα όσον αφορά την καταγραφή των εσόδων. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει χειραγώγηση στις συναλλαγές. Έτσι, η πρόληψη της απάντησης είναι ευκολότερη. Είμαστε έτοιμοι επομένω να προχωρήσουμε. Δεν χρειάζεται η λήψη και άλλων διοικητικών μέτρων. Βλέπετε τι γίνεται σε σχέση με την ε, παρέκκληση. Έχει προκύψει ότι το σύστημα μπορεί να αποτελέσει την λύση για το φαινόμενο της απάτης. Και αυτό είναι σημαντικό επιχείρημα. Επίσης, το πιλωτικό πρόγραμμα για την ε, θέση σε ισχύ αυτού του γενικευμένου συστήματος διαπιστώνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε 500.000 συναλλασσόμενους που υποχρεούνται στην απόδοση του ΦΠΑ σε πολλούς τομείς και αυτοί συμμορφώνονται με την σχετική οδηγία. Το πρώτο εξάμεινο φέτος οι φορολογούμενοι φέτος έπρεπε να καλύψουν 525 δις τσεχικές κορώνες και μιλούμε επομένως για κατόφλι 10.000 ευρώ σύμφωνα δε με υπολογισμούς μας. Αυτό σημαίνει ότι τώρα θα καλυφθούν και άλλοι 116.000 συναλλασσόμενοι. Και επίσης 53.000 περίπου νεοεισελθέντες στην αγορά συναλλασσόμενοι. Αυτοί αντιπροσωπεύουν το 10% των ε, φορολογουμένων με ΦΠΑ. Αυτά τα στοιχεία είναι επιβεβαιωμένα. είναι το σύστημα που ήδη εφαρμόζεται. Και έτσι καλύπτουμε τις συναλλαγές. Αλλά τι τις αποδείξεις για αυτές και τα σχετικά τιμολόγια. Οπότε, έτσι πιστεύουμε θα καταπολεμήσουμε την απάτη για τον ΦΠΑ. Και επομένως αυτό τελικά θα είναι ένα πλεονέκτημα για τους τίμιους συναλλασσόμενους. Έτσι αυτοί ευκολότερα θα μπορούν να εμπορεύονται και θα έχουμε λιγότερες επιλήψιμες συναλλαγές. Αυτές που αποτελούν τμήμα του φαινομένου της αλληλεγγύης απάντηση. Θα ελέγχονται καλύτερα τώρα τα τιμολόγια και έχουμε επίσης ακριβέστερα στοιχεία. Όποια κρατημέλη δεν συμφωνούν με μια τέτοια προσέγγιση δεν φύγονται από την εφαρμογή αυτής της ε, παρέκκλησης αυτού του καθεστώτος. Οπότε σας επαναλαμβάνω, η τσεχική δημοκρατία είναι έτοιμη να εφαρμόσει το εν λόγω σύστημα. Για μας είναι ένας στόχος πολύ σημαντικός. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το σύστημα να διέπεται από διαφάνεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γιάννετσεκ. Ο μιλητής μας ε, είναι ε, από το εγκληματολογικό γραφείο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε. Εμείς ε, αντιπροσωπεύουμε την αστυνομία δίωξης εγκληματικότητας και πέρα από τα φορολογικά θα κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που αφορούν γενικότερα την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Είπαμε ότι το φορολογικό ε, δίκαιο θα πρέπει να είναι πάρα πολύ στεγανό απέναντι σε καταχρήσεις, να μην ε, ανοίγει παραθυράκια και βέβαια δεν θα πρέπει να, κάνουμε, να περιοριζόμαστε μόνο σε ελέγχους, αλλά ε, και έρευνες. Ε, υπάρχει ε, εδώ ανάγκη να είναι κατάλληλο το προσωπικό για να υπάρχουν επιτυχίες στην, στις έρευνες. Σημαντική είναι η πρόληψη, θέλω να πω. Αλλά θα μιλήσω και για μέτρα, και για μέτρα κατασταλτικά. Καταρχήν, θα ήθελα να παρουσιάσω ως παράδειγμα τη γερμανική προσέγγιση, μία από τις 28 προσεγγίσεις και ε, απόψεις. Η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών και η συνεργασία είναι σημαντική και έχει να κάνει όμως και με τη δομή των ερευνητικών και διοκτικών αρχών. Εμείς ε, έχουμε 16 ε, ερευνητικέ αρχές θεωρητικά. Κάθε κρατήδιο επιλέγει τη δική του δομή. Στη Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία υπάρχουν 10 αρχές υπεύθυνε για έρευνες σε φορολογικά θέματα. Υπάρχουν και μικρότερες αρχές στα πλαίσια ενός ε, γραφείου εφορίας ε, που παρακολουθεί τα θέματα σε επιμέρους περιοχές. Έχουμε επίσης και 16 αστυνομίες δίωξης της εγκληματικότητας στην ε, Ομοσπονδιακή Γερμανία και βέβαια και σε ομοσπονδιακό επίπεδο τα τελωνία ε, και το εγκληματολογικό γραφείο υπηρεσία. Είναι σημαντική η ε, οργάνωση των αρχών αλλά από την άλλη πλευρά, ε, στην περίπτωση ας πούμε ε, αλυσιδωτών περιπτώσεων απάτης, ε, γαϊτανάκι, αυτό είναι εγκληματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες, να μπορούμε να γνωρίζουμε κάθε φορά ποιος είναι υπεύθυνο γιατί εμείς έχουμε καθορίσει ε, συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υπάρχει καλή δικτύωση, δηλαδή στις κεντρικές αρχές, στο Düsseldorf που είναι η εγκληματική υπηρεσία, ε, υπάρχουν και οι υπηρεσίες ε, που στελεχώνονται από ε, τελωνιακούς υπαλλήλους συνδέσμους και γραφεία συνδέσμους που έχουν ειδικότερες και πιο συγκεκριμένες αρμοδιότητες λείπουν κάποιες ειδικότητε βέβαια όπως παρακολούθηση ε, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Είναι σημαντικό όμως ε, να υπάρχουν για να μπορούμε να παίρνουμε στοιχεία. Και ε, στην αστυνομία δίωξη εγκληματικότητας πολλές φορές δεν υπάρχει εξειδίκευση σε θέματα νομικά και τεχνικά. Το στη Βορεια Ειρηνανία Βεσφαλία το ξέρω καλύτερα βέβαια το σύστημα, γι' αυτό αναφέρθηκα περισσότερα σε αυτό. Ε, πιστεύω, εις ό,τι αφορά κάποια αιτήματα ή υποδείξεις που μπορούμε να ε, κάνουμε, ε, ένα θέμα μεγάλο είναι η έλλειψη θεσμοθετημένης συνεργασίας. Ε, επιτυχής δηλαδή, δίωξη που θα πρέπει να ε, γίνονται πιο, πιο ε, σύντονα, συντονισμένα. Ε, εμείς έχουμε εμπειρία από εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουμε έρθει σε επαφή με το οργανωμένο έγκλημα. Πιστεύουμε ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι το οποίο εκτινάσει τις απώλειες των φόρων. Υπάρχουν ιδέες και ενδείξεις ε, ότι τα ε, κονδύλια, τα, οι φόροι που μπορούν να ε, εισπραχθούν, θα αφαιρεθούν από χέρια εγκληματιών που θα χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους άνομους σκοπούς τα, τα χρήματα αυτά. Ένα μοντέλο θα μπορούσε να είναι το σύστημα της αντιστροφής της επιβάρυνσης. Ε, αν ε, ε, θεσμοθετηθεί όμως θα πρέπει να γίνει πανευρωπαϊκά, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ, και μόνιμα, γιατί οι ε, επαγγελματίες ε, εγκληματίες θα ψάξουν και εδώ να βρουν παραθυράκια. Στην Τσεχία μπορεί... να ε, σταματήσουν να ε, δραστηριοποιούνται αν εισαχθεί ένα τέτοιο σύστημα, θα πάνε όμως σε χώρες που δεν θα το εισαγάγουν. Ε, η θεσμοθετημένη συνεργασία είναι σημαντική επίσης διότι ε, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και, τις, και αυξάνει τις επιτυχίες που δεν θα είναι τόσο πολύ το αποτέλεσμα τυχεότητας. Η, επίσης η ευθύνη, η αρμοδιότητα θα πρέπει να βρίσκεται ε, σε μία αρχή και θα πρέπει να δούμε ονομαστικά ποιος φορέας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεύθυνο για την επιτυχία ή αποτυχία στην καταπολέμηση των απατών στον τομέα του ΦΠΑ. Και στο θέμα της καταπολέμησης και άλλων μορφών εγκληματικότητας ε, είχαμε πει ότι ε, πολλές φορές δεν έχουμε να κάνουμε με εθνικές μορφές εγκληματικότητας αλλά με ευρωπαϊκή ε, εγκληματικότητα. Άρα και η λύση θα πρέπει να είναι διοκτικές αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες και τις προοπτικές συνεργασία, ε, ε, συνεργασίας ε, σε επίπεδο Europol. Η Europol έχει επιχειρησιακές αρμοδιότητες, αλλά θεωρούν ότι τα στοιχεία που παίρνουν πληροφόρηση εξακολουθεί να είναι ελλειπής και έτσι η Europol δεν στερείται ε, από τη, στερείται της δυνατότητας να ασκήσει όλες τις αρμοδιότητες ε, που έχει. Οι, ε, πολλές φορές ε, δεν δίνονται στοιχεία από φορολογικές αρχές, ε, ε, πολλές φορές παρεμποδίζονται να αποστείλουν στοιχεία, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα που δυσκολεύουν τις αναλύσεις όταν δεν υπάρχει το κόρπους των δεδομένων που απαιτείται. Ε, παρόμοια προβλήματα έχουμε και στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ε, της τραπεζικής εγκληματικότητας διασυνοριακά. Ε, θα πρέπει δηλαδή να ασχοληθούν οι αρμόδιοι υπουργοί, το Συμβούλιο Υπουργών, για να βρεθούν λύσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διευρυνθούν οι επιχειρησιακές αρμοδιότητες της Europol και να ενισχυθεί η τωρινή πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι ε, όταν είμαστε αποδυναμωμένοι σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούμε να έχουμε επιτυχίες. Ενδεχομένως θα έπρεπε να έχουμε και μια ποινική διαδικασία και ποινική δικονομία ευρωπαϊκή, σε, ευρωπαϊκό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες εκεί. Επίσης, κατά το παρελθόν, ε, είχαν ε, συμμετάσχει ε, αρμόδιοι φορείς και ιδρύματα για να επεξεργαστούν ενδεχόμενα ένα ευρωπαϊκό εταιρικό φορολογικό δίκαιο. Επίσης, αυτή η θεσμοθετημένη συνεργασία ε, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και τα θέματα ε, μετεκπαίδευσης επιμόρφωσης των αρμόδιων υπαλλήλων έρευνας και δίωξης που ακόμα είναι λύπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φίτλερ που ε, κρατήσατε και το χρόνο. Ε, πριν δώσουμε το λόγο στους θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν θέλουμε να ευχηθούμε περαστικά στο συνάδελφο ο οποίος ε, ε, ξαφνικά ασθένησε σοβαρά και ε, αντικαταστάθηκε. Παρακαλώ λοιπόν την Κομισιόν να μας παρουσιάσει τη δική της άποψη επί του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του κύριου Ραπώνη. Ε, ασθένησε σοβαρά ξαφνικά ονομάζομαι Πατρίκ Μερί, τον αντικαθιστώ σήμερα. Καταρχήν για το πρόγραμμα δράσης για το ΦΠΑ και τι πρωτοβουλίες που σκοπεύουμε να αναλάβουμε ε, για την καταπολέμηση της ε, απάτης σε θέματα ΦΠΑ. Από δική μας πλευρά, το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η απάτη ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραδεκτό το εκτιμούμε στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ ε, σε διασυνοριακές συναλλαγές συνήθως με το σύστημα του καρουζέλ. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε στο πρόγραμμα δράση μας μια ε, ενιαία ζώνη ΦΠΑ ε, δίνοντας τέλος στην προσωρινή και μεταβατική, στο προσωρινό και μεταβατικό σύστημα που ισχύει μέχρι τώρα. Έχουμε δύο δυνατότητες. Πρώτον, να αφαιρέσουμε την ε, εξαίρεση ε, των ε, διασυνοριακών ενδοκινοτικών συναλλαγών και η άλλη δυνατότητα ήταν να γενικεύσουμε το σύστημα αντίστροφης επιβάρησης, αντίστροφης επιβάρησης. Αυτές είναι οι δύο δυνατότητες, τα δύο σενάρια που έχουμε μπροστά μας και τα δύο συζητήθηκαν στην, στο Κολέγιο των Επιτρόπων και αποφασίστηκε ότι το καλύτερο θα ήταν να φορολογούνται οι συναλλαγές και όχι ε, να εξαιρεθεί όλη η αλυσίδα από το ΦΠΑ. Υπάρχουν επιχείρηματα υπέρ αυτής της αναλλακτικής. Ε, ε, πρώτον, ε, διοικητικό άχθος. Ο πρόεδρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θυμάστε τι είπε, είναι και δική μας άποψη ότι η γενίκευση της αντιστροφής της επιβάρυνσης θα αύξανε το διοικητικό άχθος. Δεύτερο επιχείρημα έχει σχέση και με άλλα που ελέγχθησαν σήμερα, με το γεγονός δηλαδή ότι μια γενίκευση της αντιστροφής της επιβάρυνσης θα δημιουργούσε καινούριου κινδύνους απάτης, ακόμα και σε επίπεδο ε, και σε άλλα κρατημέλη μάλιστα του λεχθέντος. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται επιγόντω να ληφθούν μέτρα. Γιατί το οριστικό καθεστώς α δεν θα υλοποιηθεί πολύ σύντομα. Γι' αυτό το λόγο πριν το τέλος του 2017 θέλουμε ε, να ε, έχουμε λάβει επίγοντα μέτρα. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους σε κάποια κράτη-μέλη, ονομάζονται συμβατικά, αλλά πέραν αυτών η Κομισιόν στο εκοφήν του Ιουνίου ανέλαβε να υποβάλει νομοθετική πρόταση ε, που θα υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν έναν μηχανισμό αντιστροφής επιβάρυνσης ε, σε εσωτερικές συναλλαγές πάνω από ένα όριο και ταυτόχρονα να προστατεύσουν την εσωτερική αγορά. Αυτή η πρόταση θα υποβληθεί από την Κομισιόν πριν το τέλος του χρόνου, του 2016. Τώρα, για δύο πρόστα θέματα, τα οποία ανέφεραν οι ομιλητές, να κάνουν ορισμένα σχόλια. Άλλες, χρειάζονται και άλλες πρωτοβουλίες για να η απάτη. Ε, δεν αρκεί η αλλαγή του συστήματος, χρειάζονται και άλλα πρόσθετα μέτρα, τα εντοπίσαμε στο πρόγραμμα δράσης μας για το ΦΠΑ, μάλλον είπαμε, αναφέραμε ότι θα προτείνουμε μέτρα για τη βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ ε, τελωνιακών αρχών, καθώς επίσης και μεταξύ ε, τελωνίων και ε, αστυνομίας. Έχουμε ε, επίσης ε, πρόταση για τροποποίηση των ρυθμίσεων ε, που αφορούν και το Eurofisc και γενικότερα την διοικητική ε, συνεργασία. Ε, αυτές θα υποβληθούμε στο 2017. Τέλος σχόλιο, τελευταίο σχόλιο που έχει σχέση με ένα συγκεκριμένο τομέα στον οποίο η απάτη είναι ιδιαίτερα σημαντική που είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σκοπεύουμε να υποβάλουμε μέχρι το τέλος του χρόνου πρόταση για να ε, διευρύνουμε τον ε, μηχανισμό του mini stop shop, one stop shop, ε, ενώ ταυτόχρονα θα ακυρώσουμε ε, την εξαίρεση για μικρές εισαγωγές ε, και θα πάρουμε και μέτρα διευκόλυνσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος αυτού του πακέτου θα είναι η απλοποίηση του διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα η καταπολέμηση της απάτης. Στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου οι απώλειες ΦΠΑ εκτιμώνται να ανέρχονται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και εκτιμάται ότι θα φτάσουν στο 7 δισεκατομμύρια μέχρι το 2021. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και για το ότι πρόθεσμα ε, κλείθητε να αντικαταστήσετε τον ε, ε, προ... προϊστάμενό σας. Ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα. Ο σκιώδης συζητητής μας ζητεί να τον συγχωρήσετε, διακόπτη η κυρία Μπέρες, Κύριε Τζάνη δεν μπόρεσε να παραστεί και ζήτησε να τον αντικαταστήσω για ε, αυτή την πρώτη σειρά των ερωτήσεων. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε όλους τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν από την άλλη μεριά. Δεν είμαι τόσο σίγουρη ε, τώρα τι πρόκειται. Πρόκειται για λομπίστε ή εμπειρογνώμονε, Δεν είμαι σίγουρη. Εξαρτάται ε, περίπτωση, αλλά ε, τέλος πάντων στην ε, ακρόαση αυτό δεν προκύπτει σαφώς και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε το τι λέει ο καθένα με τις ερωτήσεις. Η αυτορευστοποίηση είναι πιο σημαντική ίσως, το σημαντικό και τελικά οι συνάδελφοι που οποίοι από τον τελευταίο κρίκο της Αλυσίδα για τη φορολόγηση ε, νομίζω ότι εμφανίζεται εδώ πέρα κάποια αντίφαση σε σχέση με την αρχή της καταπολέμησης της ε, πάντης. Άκουσα ότι είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει επιγόντως να ληφθούν ε, μέτρα. Ναι, ε, αυτό αφορά την καταπολέμηση της απάτης. Για πάντως, είναι ζημιογόνο το να κάνουμε κάτι το οποίο θα χτυπούσε όλους τους κρίκους της αλυσίδας που τόσο καιρό κοπιάσαμε για να στήσουμε για όλη την διαδρομή που οδηγεί στην επιβάλληση με το ΦΠΑ χωρίς να έχουμε καμία απόδειξη, καμία εγγύηση ότι ό,τι κάνουμε θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ε, απάτης. Αντίθετα, έχουμε και το ρίσκο του να αυξηθεί η απάτη. Τώρα, όσον αφορά αυτά τα trusted deals που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε ε, να εφαρμόσουμε, αυτό θα αφορά και θα είναι πιο αποτελεσματικό με τις διασυνοριακές συναλλαχές και να έχουμε μία βαθμιαία εφαρμογή οριστικού συστήματος και επίσης να έχουμε μεταβολή του τόπου ίσπραξης του φόρου. Επιτρέψατε μου πρόεδρε, έχω και κάποιες ερωτήσεις πρώτα-πρώτα θα έχουμε κάποια λίστα, κάποιο κατάλογο ε, για κάποιους μειωμένους συντελεστές, το οποίο θα επικαιροποιείται κάθε τόσο από πλευρά των κρατών μελών. Έτσι θα έχουμε ε, κάποιο είδους εξαιρέσεις, κάποιες παρεκκλήσεις με μικρότερο συντελεστή. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας μιλά για αποτελεσματική καταπολέμηση της ε, απάτης. Δηλαδή να ενισχυθεί ο, να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του εισαγγελέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ζητηθεί και από την ε, Νομική Επιτροπή. Να μας πούν τι πρεσβεύουν σε αυτό οι καλεσμένοι μας. Τώρα κάτι άλλο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια συγκεκριμένη περίπτωση απάντηση. Έχουμε ασχοληθεί με αυτή την περίπτωση και ήδη έχω απευθυνθεί στην Επιτροπή κ. Βέσταγκερ, αλλά και στον Επίτροπο κ. Μοσκοβησί και αφορά την απάτη για τον ΦΠΑ όσον αφορά τους ε, κτηνοτρόφους που ασχολούνται με το χείριο κρέας. Γιατί εκεί υπάρχει κάποια ε, διάκριση και ο ε, παραγωγός δεν επιβαρύνεται. Θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ισχύει. Ευχαριστώ. Κύριε Σλόξ, ευχαριστώ πολύ. Στα γερμανικά θα μιλήσω. Στις ερωτήσεις μου θα εστιάσω στη δυνατότητα συστήματος αντιστροφής της επιβάρυνσης. Είπατε, είπε η Κομισιόν, και νομίζω και ο πρώτος ομιλητής, ότι το σύστημα αντιστροφής της επιβάρυνσης οδηγεί σε αυξημένες διοικητικές δαπάνες. Δεν κατάλαβα γιατί το reverse charge θα στοιχίζει περισσότερο από το τωρινό σύστημα χρεώσεων επιβαρύνσεων. Αυτό που δεν αξιολογήθηκε όπως πρέπει είναι το γεγονός ότι η αντιστροφή της επιβάρυνσης είναι πολύ λιγότερο επαχθές ε, για τους εμπλεκομένους. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να παίξει ρόλο κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Επίσης, αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Γιάννετσεκ είπε ότι υπάρχει και πρακτική εμπειρία η οποία δείχνει ότι η διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης ε, είναι πιο ανθεκτικό από το την κανονική επιβάρυνση είναι πιο ανθεκτικό στις απάτες. Αν ισχύει ότι μειώνονται στην Τσεχία οι περιπτώσεις απάτης με το ΦΠΑ, τότε αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται τα έσοδα από τους φόρους. Ε, μήπως μπορεί να μας πει σε ποιο ποσοστά μειώθηκε η εγκληματικότητα σε αυτό το τομέα μετά την εφαρμογή του reverse charge. γιατί ενδεχομένως αυτό θα βοηθήσει ε, να αλλάξουν και τα άλλα συστήματα. Επίσης, καταλαβαίνω βεβαίως απόλυτα την παρατήρηση που έγινε σχετικά με την ενδεχόμενα προσωρινή εφαρμογή αυτού του συστήματος, πράγμα που θα οδηγήσει σε ανασφάλεια, βεβαιότητα, ε, δεν ε, αν είναι προσωρινό ή αν ισχύσει σε ορισμένους μονοκλάδους αυτό δεν θα, θα δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά η πρόταση για γενικότερη αντιστροφή της επιβάρυνσης ε, συζητείται ακόμη, δεν έχει ε, απορριφθεί αν συνεργαστούν όλα τα κράτη. Τώρα, αν δεν συνεργαστούν όλα τα κράτη, γίνεται να υπάρχει αντιστροφή της επιβάρυνσης σε κάποια κράτη-μέλη μόνο αφού θα είναι ας πούμε, κυρίαρχη απόφαση των φορολογικών αρχών αυτών των κρατών μελών, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη δεν θα ληφθεί σχετική απόφαση. Αυτή η ερώτηση αφορά όλους τους εμπειρογνώμονες. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα, όντως, αν κάποια κράτη-μέλη ενεργοποιήσουν ένα σύστημα αντιστροφής επιβάρυνση και άλλοι όχι. Στο βαθμό που υπάρχει η αρχή της χώρας προορισμού, ε, σε διασυνοριακές συναλλαγές δεν υπάρχει ε, αντίφαση μεταξύ των δύο συστημάτων, δηλαδή reverse charge σε ένα κράτος μέλος και όχι σε ένα άλλος. Δηλαδή, αν υπάρχει πρόβλημα, δεν θα ήθελα να μου, να μου εξηγήσετε τι πρόβλημα θα προκύψει σε μια τέτοια περίπτωση. Ο κ. Γιάσεκ για τους φιλελεύθερους. Θα ήθελα και εγώ μια απάντηση στι ερωτήσει του κ. ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το διοικητικό βάρος. Θα μπορούσαν οι ομιλητές να είναι λίγο πιο σαφείς σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, πόσο θα είναι το διοικητικό βάρος και μήπως θα είναι μάλιστα και υπερβολικά βαρύ, σε υπερβολικά μεγάλο σε σχέση με το στόχο και τα ωφέλη. Δεύτερον, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για το θέμα της νομικής αβεβαιότητας Επίσης το ελεγκτικό συνέδριο, αν κατάλαβα καλά, είπε το σύστημα είναι καλό και το πρόβλημα είναι η αδυναμία σε του. Ιδιαίτερα συγκεκριμένα έξι κράτη-μέλη. Αν δούμε όμως το επίπεδο της απάτης, ε, διαψεύδεται ε, αυτή η άποψη. Δηλαδή θα πρέπει και το ίδιο το σύστημα να έχει προβλήματα, όχι μόνο η εφαρμογή του. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις απάτες τύπου καρουζέλ και απουσία συναλλασσόμενου. Ασφαλώς και χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά δεν νομίζω ότι θα αρκεί, διότι ε, οι, αυτοί που εκμεταλλεύονται τις ανανεμίες συστήματος ε, είναι ευέλικτοι, μετακινούνται από κράτος σε κράτος, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Αν έχετε βέβαια κάποια ιδέα, πολύ ευχαριστώ να την ακούσω. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε το πιλωτικό project με την αντιστροφή της επιβάρυνσης ε, γιατί αλλιώς ε, δεν θα, θα κολλήσουμε. Θα κολλήσουμε. Η κυρία Ντανιέλ για την αριστερά, για τους, η κυρία Μόνης Καρτάτο και για ε, τους πράσινους, ο κύριος Τσάνη για την FDD. Αλλά κανείς δεν είναι εδώ. Θα εκπροσωπηθούν από άλλον. Όχι. Εντάξει, κυρία Κάπελη, ΕΝΕΦ. Ευχαριστώ. Προχωρήσαμε πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε πολύ τους κυρίους για τις παρατηρήσεις τους. Αυτά που μας είπατε μας βοηθούν να προχωρήσουμε. Αποκρισταλώνονται κάποια θέματα με παραδείγματα που είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε το θέμα των ελληπών πληροφοριών, ανταλλαγών πληροφοριών ή την έλλειψη τέτοιων πληροφοριών ε, και η Όλαφ και η Europol και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, δεν έχουν ε, πρόσβαση στα δεδομένα των κρατών μελών πάντοτε και ακούσαμε από την αστυνομία ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υφίσταται ανταλλαγή δεδομένων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να, να ακολουθήσουμε το ελεγκτικό ε, συνέδριο και να βρούμε μία online εφαρμογή για τον ΦΠΑ. Είναι πολύ σωστή η πρόταση αυτή. Με εντυπωσίασε επίσης ο μεγάλος αριθμός ε, της μείωσης των απατών στην Τσεχία. Κάτι είπατε για 98% που μου φαίνεται ε, πολύ εντυπωσιακό. Και οπωσδήποτε ε, και στο ΕΚΟΦΗΝ οι υπουργοί ε, θα προβλέψουν τη δυνατότητα ενό συστήματος ε, ε, reverse charge, γιατί 98% ποσοστό επιτυχίας είναι πάρα πολύ ψηλό. Και εγώ ήμουν στην αρχή επιφυλακτική, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ και την πρόσθετη γραφειοκρατία, αλλά μου φαίνεται ότι αφού είναι τόσο υψηλή η επιτυχία, 98%, ε, πρέπει να του δώσουμε μια ευκαιρία αυτού του συστήματος. Ε, το, το τρίτο που τόνισε ο κύριος Φίτλερ, ε, δίωξη στα χέρια ενός καθορισμένου ονομαστικά και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας βυσής μας είπατε για τη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, μπορούμε να τα δούμε και εμείς ε, αυτά, να κρίνουμε δηλαδή ε, πώς λειτουργεί το μοντέλο και να προτείνουμε εντατικοποιημένη και θεσμοθετημένη ε, συνεργασία με βάση αυτό το παράδειγμα. Η απάτη στον ΦΠΑ είναι τεράστιο πρόβλημα για τα κράτη-μέλη. Ακούσαμε μεταξύ 50 δις μέχρι 170 δις το χρόνο που χάνονται. Τα κράτη-μέλη λοιπόν ενδιαφέρονται πάρα πολύ όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρουν κανόνες για να μειωθεί το πρόβλημα. Και ελπίζομαι ότι μπορεί να είναι ένα καλό μέσο η αντιστροφή της επιβάρυνσης και σίγουρα η καλύτερη ε, ενημέρωση και η ανταλλαγή πληροφοριών ε, θα αναβαθμιστούν. Ε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα μετά από προσωρινά μέτρα να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα αποφασιστικά βήματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάπελ. Τώρα στα πλαίσια του Catch the Eye τρεις ομιλητές ε, ζήτησαν το λόγο. Για ένα λεπτό. Κύριος Ντενανό. να σας μιλήσω για το ότι εδώ και 20 χρόνια υπάρχει κάποιος κλάδος που αναπτύσσεται. Πρόκειται για τα άλογα. Για γεωργικές χρήσεις, αλλά και αθλητικές, αλλά και ψυχαγωγία. Η νομοθεσία οδήγησε όμως σε κάμψη του κλάδου για την λόγους αύξησης του συντελεστή. Τώρα αντιμετωπίζει ο κλάδος αυξημένες δυσκολίες, όπως και όλη η Γεωργία, μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία. Θα πρέπει να αποκρισταλωθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα ΦΠΑ. Και με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την τροποποίηση της σχετικής οδηγίας, που θα πρέπει να καλύψει και την ρύθμιση αυτού του προβλήματος και τα δέκρατη μέλη να μπορούν να επιλέξουν ποιο συντελεστής θα εφαρμόζεται για κάθε δραστηριότητα. Ευχαριστώ κύριε Νίδερ Μάιερ. είμαι σύντομο. Πρώτον, να αναζητούμε ευρωπαϊκή λύση, γιατί η λειτουργία τη εσωτερική αγορά είναι από τα βασικά του τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με του ομιλητέ. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε καλύτερα το καινούριο βήμα, αν δεν το μετρήσουμε, αν δεν το σταθμίσουμε, δεν μπορούμε να μετρήσουμε και την πρόοδο. Επίσης, συμφωνώ ότι έχουμε δύο εναλλαγές. Πρώτον, μια ενιαία ε, ζώνη ΦΠΑ, παρόμοια με το σημερινό σύστημα ε, και λύνει το διασυνοριακό πρόβλημα. Γιατί τα περισσότερε απάτε καρουζέλ σχετίζονται με διασυνοριακές συναλλαγέ. Ε, και θα νομίζω λοιπόν ότι η αντί για αντιστροφή της επιβάρυνσης ε, η άλλη ανατική λύση αφορά την αναστολή ε, ΦΠΑ. Αυτό όμως θα δημιούργησε περισσότερα προβλήματα. Ε, αν δηλαδή η αντιστροφή της επιβάρυνσης ε, εφαρμοστεί μόνο σε ορισμένα ε, σημεία, σε ορισμένους τομείς κλπ, ε, τότε θα δημιουργηθούν περισσότερες, περισσότερα προβλήματα στην ανάκτηση, στην επιστροφή του ΦΠΑ. οπότε πρέπει να εξετάσουμε πολύ καλά τα πράγματα και να μην κάνουμε πειράματα εντωμεταξύ. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, και εσά και του προσκεκλημένου. Θέλω να σα πω το εξή, ότι φέτο το ελεγκτικό συνέδριο σκέφτηκε με την Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Λετωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Διεπίστωσαν ότι στα περισσότερα από αυτά τα κρατη δεν υπήρχαν αποτελεσματικοί έλεγχοι ε, ε συναλλαγέ. Ε, δεν υπήρχε διασταύρωση των στοιχείων των τελωνίων και υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά το, την πληρότητα, το, το, το timing ε, και την ε, ακρίβεια. Και υπήρχαν επίσης και κάποιες επικαλύψεις μεταξύ του έργου των διοικητικών αρχών, των διοικητικών αρχών και δικαστικών. Και αυτά τα λέει και λίγο συνέδριο ότι σε κάποια περίπτωση ένα κράτος μέλος υπήρχε λάθος αριθμός ΦΠΑ και αυτό διαβιβάστηκε από κάποιο κράτος μέλος ε, δύο χρόνια αργότερα. Και ούτε η Europol, ούτε η Όλαφ έχουν προσβασιμότητα σε στοιχεία κάποιου κράτους μέλους όσον αφορά τα δίκτυα και την πολέμηση της ε, απάτης, αλλά και την ανταλλαγή των σχετικών στοιχείων. Μπορείτε να μας ενημερώσετε. Έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις σχετικά με αυτά, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αργών από τον Μάρτιο του 2016. Το 2011 είπαμε ότι πρέπει να αναθεώρηση το άρθρο 42 για την τελειωνική διαδικασία όσον αφορά την πρώτη χώρα που θα εισαχθεί κάτι. Δεν έκανε τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χάνουμε 40 έως 60 δις όσον αφορά μη εισπρατώμενο ΦΠΑ. Πώς είναι δυνατόν να καταφέρουμε να αναθεωρήσουμε, να τροποποιήσουμε τέλο πάντων τον λόγο άρθρο. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τα κόμματα, κάναμε και τη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ. Ο λόγος του εμπειρογνώμονες για πέντε λεπτά, ο κύριος Καρακατσάνης. Καταρχήν, ευχαριστώ. Okay. Ε, ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Καταρχήν, ο πρόεδρος μου είχε υποβάλει δύο ερωτήματα στην αρχή τι, ποια θεωρούμε ότι είναι τα πιο επίγοντα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Αυτό έχει σχετίζεται με το τελευταίο σχόλιο που έγινε. Και δεύτερον, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την καταπολέμηση απάτης. Το είπα και στην αρχή. Ε, μίλησε για τα νούμερα. Ακόμα και σήμερα εδώ ε, από έναν από τους ομιλητές ε, μιλήσαμε για τις διαφορές στην εφαρμογή του συστήματος. Ε, πέραν του γεγονότος ότι περιλαμβάνονται απάτες και εσωτερικές και διασυνοριακές, περιλαμβάνονται όμως και άλλες, άλλα συστήματα όπως νόμιμη αποφυγή, φοροαποφυγή δηλαδή του ΦΠΑ, με πολλούς τρόπους. Το χάσμα αυτό σχετίζεται επίσης και με την ε, μαύρη οικονομία ε, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο, στην υπολογισμό του ΑΕΠ. Οπότε ε, πρέπει να ξέρουμε πώς να μετρήσουμε πρώτα την απάτη ΦΠΑ. Αν ξέρουμε πώς να τη μετρήσουμε μπορεί να φτάσουμε στα 40 ή 60 δισεκατομμύρια. Στην μελέτη την οποία χρησιμοποίησε η Κομισιόν ε, δεν, δεν, τα κριτήρια που ελέγχθησαν υπόψη δεν είναι ακριβή, δεν είναι ασφαλή. Μπορώ να σας το εξηγήσω με, με λεπτομέρεια. Ε, δεν είναι σαφές ότι αυτά τα νούμερα είναι ακριβή και αξιόπιστα και, αυτό, και πρέπει να ξεκινήσουμε με καλύτερες μετρήσεις λοιπόν. Τώρα σε ό,τι αφορά τα επίγοντα μέτρα με το ισχύον σύστημα είδαμε στο ισχυρό σύστημα είδαμε ότι το σύστημα αυτό είναι βάσιμο, είναι ε, ασφαλές, ε, αλλά δεν εφαρμόζεται σωστά. Πώς θα εφαρμοστεί σωστότερα, είπαμε, κάναμε συστάσεις. Μεταξύ αυτών και την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ τελωνίων και ε, φορολογικών αρχών. Σύσταση την οποία δεν δέχτηκε η Κομισιόν. Οι περισσότερες συστάσεις μας όμως ελήφθησαν υπόψη. Και το βλέπουμε αυτό σιγά σιγά. Και κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά την αντιστροφή της επιβάρυνσης. Τι είπαμε εμείς στην έκθεσή μας. Παράγραφοι 87 και 88. Είπαμε ότι δεν συμφωνούμε με την Τσεχική Δημοκρατία. Λέμε ότι είναι χρήσιμο εργαλείο που δεν χρησιμοποιείται συχνά. Εμεί θεωρούμε ότι η αντιστροφή τη επιβάρηση είναι χρήσιμο εργαλείο όταν εφαρμόζεται από όλα τα κράτη-μέλη, ε, ιδιαίτερα σε ε, τομεί κινδύνου. Σε μία έρευνα που κάναμε, η Τσεχική Δημοκρατία είναι το μόνο από αυτά τα κράτη-μέλη που ρωτήσαμε που είναι υπέρ τη γενίκευση της αντιστροφή τη Το πρόβλημα με την αντιστροφή τη επιβάρυνση, όπω είπε και η Κομισιόν, είναι ότι μετακινεί την απάτη από άλλα στάδια στον, στο τελικό στάδιο της λιανικής πώληση. Το λέμε στην παράγραφο 89 της έκθεσή μας. Δεν θεωρούμε ότι θα είναι αποτελεσματικό αυτό το σύστημα κατά πολέμηση απάτης, γιατί στην, ε, στο τελευταίο στάδιο της λιανικής εκεί η κίνδυνη είναι ακόμα υψηλότερη για απάτη. Οπότε πιθανώς να επιδεινωθεί η κατάσταση αντί να βελτιωθεί, αν γενικευθεί η αντιστροφή της επιβάρησης. Το ό,τι αφορά το ύψος της απάτης είπαμε ότι το σύστημα είναι ε, ε πλήρες. Ε, έχει προβλήματα εφαρμογής. Έχουμε παραδείγματα. Έχουμε προβλήματα τα οποία όμως δεν είναι ξεπεραστα Δύο κρατημέλη βελτίωσαν δραματικά την εισπράξη του ΦΠΑ με τη λήψη ειδικών μέτρων. Και η Κομισιόν θα μπορούσε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές να τις ε, προωθήσει μέσω των συστημάτων που ήδη υπάρχουν. Υπάρχουν συστήματα ανταλλαγή πληροφοριών και των πρακτικών. Τώρα, Εμεί δεν είπα ότι δεν είχαμε πρόσβαση στα αρχεία, δεν είχαμε τέτοιου είδου προβλήματα. Είπα ότι η Europol και η Όλαφ έχουν κάποια θέματα πρόσβαση. και νομίζω ότι το ανέφερε και ένα άλλο από τους ομιλητέ. Χαίρομαι που η Κομισιόν παίρνει μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Αυτά. Ähm, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χίμερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω για δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα για την αντιστροφή της επιβάρυνσης. Η, ΜΜΕ τι κάνουν. Δεν έχουμε τώρα ούτε σε ένα κράτος μέλος που να μπορούν οι ΜΜΕ να μπορούν να έχουν αξιόπιστες πληροφορίες από πλευράς φορολογικών αρχών. Γιατί εάν δεν υπάρχει ο πελάτης, να ο πελάτης είναι ο τελικός καταναλωτής, τότε η ΜΜΕ στέλνει το τιμολόγιο χωρίς τον ΦΠΑ. Το υποβάλλει και κατόπιν γίνεται η αφαίρεση, η έκπτωση και επιστρέφονται τα χρήματα αν έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ. Και αυτό είναι που καίει τι ΜΜΕ. Άπαξ και τα ΜΜΕ δεν έχουν αξιόπιστα στοιχεία στα οποία να μπορούν να στηριχτούν τότε. Το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο. Κάτι άλλο τώρα για το άχθο. Όπω είπατε, εάν έχουμε προσωρινή θέσπιση του συστήματο και μόνο για κάποιου τομεί, κάποιου κλάδου ή μόνο για κάποιε εταιρείε τότε θα πρέπει οι ΜΜΕ να αποφασίσει τι ισχύει. Ισχύει η συνείδηση επιβάρυνση ή η αντιστροφή. Οπότε και χρειάζεται ε, να κάνει πάρα πολλά γραφειοκρατικά εταιρεία και μιλάμε για δύο-τρία χρόνια, τότε θα πρέπει να, ε, να ξαναγυρίσει το παλαιότερο σύστημα όταν σταματήσει η προσωρινή εφαρμογή. Άρα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα κατημέρια το σύστημα. Όμω τότε να γίνουν τα προβλήματα που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο συνέδρος από το Ελληνικό Συνέδριο. Ότι δηλαδή μετακυλεί το κίνδυνο στην τελική φάση. Έχει δίκιο επομένω στην προκειμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά πρέπει να υπάρχει ενιαία φορολογική πολιτική, ενιαία εφαρμογή. Κάτι άλλο τώρα που θέλω να σα πω είναι όσον αφορά τον κατάλογο για το που υπάρχει μειωμένο συντηλεστή. Εάν εφαρμόσουμε την αρχή του προορισμού και πάλι θα έχουμε κάποια κρατημέλη τα οποία θα έχουν μειωμένου τελεστές για να ελκύσουν καταναλωτέ από το εξωτερικό. Και ας πούμε, θα πηγαίνουν υπερβολικά πολύ, να πηγαίνουν στο Λουξεμβούργο α πούμε γιατί θα έχει μειωμένο συντελεστή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν θα υπάρξει σημαντική επίπτωση εις ε, την εσωτερική αγορά, εάν μπορούν ελεύθερα τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν τι συντελεστή θα εφαρμόσουν, πού θα έχουν ε, επομένως ε, μειωμένο συντελεστή, πού θα εφαρμόσουν κάποιες παρεκκλήσεις. Αυτό είναι κατά της ενιαίας αγοράς. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. το λόγο στον κύριο Γιάννετσεκ. πρώτα πρώτα να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κύριος Καρακατσάνης που είπε για τη δική μας πρόταση υπέρ αυτού του καινούργιου στήματος. Όχι, υπάρχουν και άλλα κρατημέλη που μας ε, υποστηρίζουν. Έχουμε πέντε κρατημέλη που συνεφώνησαν και μαζί με εμάς υπέβαλαν το σχετικό αίτημα. Άρα δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που είπατε. Επίσης είπατε ότι δεν θα αποδώσει το σύστημα γιατί θα μετακυλιστεί. Η απάτη θα μετατεθεί σε άλλο κράτος μέλος. Μα αυτό σημαίνει ότι το σύστημα αποδίδει. Γιατί αν είναι αυτή η αντίδραση, τότε αποδίδει η αντιστροφή της επιβάρυνσης. Και υπάρχει ο κίνδυνος να πάει, είπατε, η απάτη στο τελικό στάδιο. Πάντως η εμπειρία μας έχει δείξει ότι είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσει κανείς την απάντηση στο τελικό στάδιο παρά αλλού στην αλυσίδα. Μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια τα οποία καταβάλλονται για συναλλαγές διασυνοριακές. Και αν ε, κάποιος δεν έχει δηλωθεί ως βασικός εταίρος μιας ΕΠΕ, τότε δεν μπορείτε να ελέγξετε. Και θα υπάρχει πρόβλημα στο τελικό στάδιο της συναλλαγής, γιατί τότε αγαθά και υπηρεσίες θα είναι αντικείμενο συναλλαγών στην αγορά και ο καταναλωτής θα αγοράζει από κατηγορία, από σύνολο από εταιρεία που ακολουθεί επιλήψιμες πρακτικές. Όχι, δεν θέλω να πω ότι δεν μας αρέσει το σύστημα του One Stop Shop, αλλά το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει αυτό στην Ευρώπη. Και την αντιστροφή της επιβάρυνσης, όμως ξέρω πώς θα λειτουργήσει που μπορεί αυτό να γίνει άμεσα στην τσεχική δημοκρατία. Πώς όμως θα λειτουργήσει το One Stop Shop, ε, αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Εσείς θέλετε ένα σύστημα, οπότε θα εφαρμόζεται, ε, θα επιβάλλεται αυτόν τον φόρο για διασυνορικές συναλλαγές. Πώς όμως θα έχουμε την επιστροφή του φόρου όταν έχουμε δύο εταιρείε που έχουν καταβάλει σε διασυνορική συναλλαγή τον φόρο. Έτσι θα έπρεπε να έχουμε κάποια συνολική, απόλυτη συνεργασία των φορολογικών αρχών. Από πού θα γίνει η επιστροφή του φόρου, θα γίνεται η καθάριση. Δεν ξέρουμε. Τι θα προκύψει με ένα τέτοιο σύστημα. Οπότε περιμένουμε να μας τα αναλύσετε και έτσι να αποδείξετε ότι είναι καλύτερο το One Stop Shop. Δεν νομίζουμε εμείς ότι έτσι θα καταπολεμηθεί η απάτη. Πιστεύουμε ότι η απάτη θα συνεχίσει να υπάρχει όσο υπάρχουν φόροι που επιβάλλονται. Να γίνει όμως μία ανάλυση για να δούμε πώς είναι δυνατόν να κινηθεί μεταξύ περισσότερων κρατών μελών η φοροαποφυγή. Εμείς έχουμε προβληματιστεί πάνω σε αυτό και θεωρούμε ότι αν εφαρμοστεί ένα πιλωτικό πρόγραμμα τότε θα έχουμε μια ιδέα για το πόσο χρήσιμο είναι το σύστημα τη ανεσπροφής επιβάρυνσης για να αποτεμήσουμε το πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά την απλούστευση. Έχουμε προσπαθήσει να αναλύσουμε τι γίνεται με το διοικητικό άκθος. Δεν νομίζουμε ότι η απλούστευση θα βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση για το διοικητικό άρθρος. Η ισχύουσα οδηγία επιτρέπει την εφαρμογή τη αντιστροφή επιβάλλησης για συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορεύματα. Πάντω είναι δύσκολο κάθε φορά να κρίνεται εάν κάποιο προϊόν ή όχι, ε, εάν κάποιο προϊόν ή κάποιο εμπόρευμα υπάρχει στη ρύθμιση του κατοφλίου των 10.000 ευρώ. Κατά αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται κάποιοι κίνδυνοι. σταθμίζονται τέλος πάντων. Και τη σήμερα ημέρα ακόμα υπάρχουν πολλά φαινόμενα διοικητικού άχθους γιατί το σύστημα είναι υπερβολικά περίπλοκο. Μια που εφαρμόζεται το σύστημα ανά επίπεδο αναφάση συναλλαγής. Έτσι, οι υπόχρεοι φόρο δεν έχουν ασφάλεια δικαίου. Θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι σημαντική συναλλαγή και τι είναι λιγότερο σημαντική συναλλαγή. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, μιλήσαμε για την μείωση της απάντηση κατά 98%. Αυτά. Also wenn Sie, wenn Sie es uns schnell noch sagen könnten, dann wären wir alle da. Πείτε mal, και αυτό για να έχουμε πλήρη εικόνα. Καλά. Λέει ο Κάποιοι εξεπλάγησαν με το ποσοστό θα της μείωση της απάντησης κατά 98%. Ναι, σύμφωνα αυτό. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Ε, αυτό γίνεται σε ορισμένε περιπτώσεις και αφορά συγκεκριμένα προϊόντα, με εμπορεύματα. Είπατε ότι αν εφαρμοστεί κάπου αυτό, μετά η απάτη θα πάει αλλού. Όχι, δεν είναι έτσι. Σταμάτησε έτσι η αλυσιδωτή απάτη. Και όσον αφορά τώρα τι δημοσιονομικέ συνέπειε, ε, και την ίσπραξη των φόρων. Όχι, δεν είχαμε παραπάνω φόρο ο οποίο εισεπράχθη γιατί πήγε απάτη σε άλλο εμπόρευμα. Όμως στην περίπτωση αυτής της ε, απάτης θέλουμε να υπάρξει ένα καινούργιο καθεστώς ώστε να εντοπίσουμε τα σχετικά την, την μέσω αυτών των τιμολογιών. Ευχαριστώ. Λίγα έχουν μείνει να απαντηθούν. Η πρώτη ερώτηση ήταν προς ε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή για ενημέρωση, ανταλλαγή πληροφοριών, ποιων πληροφοριών συγκεκριμένα. Η εξίσωση για μας σε αυτές τις περιπτώσεις εγκληματικότητας είναι ότι πρέπει να θέσουμε το ερώτημα πώς θα καταπολεμήσουν την ευρωπαϊκή εγκληματικότητα και αν μπορεί να υπάρχει ιδέα ότι τέτοιες μορφές μπορεί να επιλύονται μόνο από τις εθνικές αρχές. Γιατί ε, για κάθε τηλεφωνικό αριθμό, αριθμό τηλεφώνου που ερευνούμε θα πρέπει να ε, προχωράμε σε 11 ε, μέτρα έτοιμα δικαστικής, έτοιμα συνδρομής ε, και όλα αυτά είναι πολύ επαχθείς και ε, χρονοβόρες διαδικασίες. Κάθε μέρα έτσι πρέπει να δουλεύουμε. Και πιστεύω ότι έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα της ασφάλειας, εσωτερικής ασφάλειας, και εδώ μπαίνει, συγκαταλέγεται και αυτό το θέμα της εγκληματικότητας, οικονομική εγκληματικότητα, που είναι στενά συνειφασμένη με, με το οργανωμένο έγκλημα, αυτό είναι πολύ σημαντικό και κομμάτια του οργανωμένου εγκλήματος ε, ε, δυναμώνουν με κάθε δισεκατομμύριο που χάνεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ε, ανησυχεί τους πολίτες συνεχώς. Και οι πολίτες βλέπουν ότι έχουμε 28 διαφορετικές διαδικασίες και για κάθε ε, αριθμό τηλεφώνου που θέλουμε να ε, ακούσουμε πρέπει να ε, υποβάλλουμε αίτημα συνδρομής. Ε, πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας καλύτερος τρόπος που να αξιοποιεί και το χώρο Σέγγεν. Όπως δημιουργήσαμε τον, το, το Σέγγεν, έτσι θα προχωρήσουμε και εδώ. Δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω και πραγματικά σας παροτρύνω και σε αυτούς τους τομείς της εγκληματικότητας, πέρα από τρομοκρατία που κάναμε παρόμοια, να μας υποστηρίξετε γιατί κατεπηγόντως θέλουμε να κάνουμε πιο αποφασιστικά βήματα για περισσότερη Ευρώπη στον τομέα της δίωξης. Θέλουμε χώρο ερευνών και δίωξης ευρωπαϊκό για την καταπολέμηση αυτής, αυτών των μορφών απάτης. Ε, γι' αυτό είναι σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε αποτελέσματα που να ανταποκρίνονται στις ε, ε, ε, ε προσδοκίες μας. Ε, και η Όλαφ, η Europol δεν μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όπως είναι διαμορφωμένα σήμερα. δεν είναι όπως ο Αμερικανικός FBI το, το FBI. Ε, ο υπεύθυνο ε, των ερευνών που εξετάζει μια υπόθεση θα πρέπει να έχει άμεση, σε μια χώρα μέλος θα πρέπει να ε, έχει άμεση πρόσβαση σε ευρωπαϊκά δεδομένα και ευρωπαϊκές αρχές και φορείς. Θα πρέπει να φροντίσουν λοιπόν οι αρμόδιοι ε, υπουργοί ε, να λάβουν αποφάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών που θα βοηθήσουν ε, να μειωθεί ε, το, το, το άχθος κάθε υπαλλήλου, δημιουργώντας τις κατάλληλες δομές. Και έτσι θα μπορούν να λαμβάνονται ευκολότερα και πολιτικές αποφάσεις. Και για να πάω στον κύριο Λούκε, γιατί η συζήτηση που άκουσα ε, κρατάει εδώ και 15 χρόνια. Δηλαδή reverse charge και ποια κράτη θα συμμετέχουν και ποια κράτη δεν θέλουν να συμμετέχουν. Ε, για να απαντήσω λοιπόν, ε, ε, εμείς ε, αντιμετωπίζουμε ε, επαγγελματίες απατεώνες και σαφώς οι άνθρωποι αυτοί θα επιλέξουν τις, ε, τα προσφορότερα καθεστώτα ε, για να ε, δραστηριοποιηθούν. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ευρωπαϊκή ενιαία προσέγγιση στα πλαίσια της πρόληψης. Το θέλουμε ή θα αφήνουμε και στο μέλλον παραθυράκια που θα τα αξιοποιούν οι ίδιοι οι εγκληματίες οι οργανωμένοι. Ευχαριστούμε πολύ και που τηρήσατε το χρόνο σας η Κομισιόν. Πολλά ελέγχθησαν για το θέμα, αλλά εγώ θα απαντήσω για τη διαδικασία εισαγωγής 42. Ε, Μας ρωτήσανε τι κάνουμε. Ε, καταρχήν να σας πω το εξής, ότι η νομοθεσία ενισχύθηκε πολύ πρόσφατα και αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Η ομάδα εργασία όμως εργάζεται και για να υποβάλει στάση για το πώς θα βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στι εθνικές, φορολογικέ και τελωνιακέ αρχές. Με αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων του ΦΠΑ στην ε, διαδικασία της εισαγωγή. Η ενιαία ζώνη ΦΠΑ, την οποία προτείνουμε, έχει ως στόχο ακριβώς να ε, καταργηθεί ο λόγος για την ύπαρξη διαδικασία 42.00. Ο λόγος αυτός ήταν ότι ε, έχουμε μια απαλλασσόμενη εισαγωγή που ακολουθείται από μια απαλλασσόμενη ενδοκινοτική διακίνηση. Οπότε με τον τρόπο που με τη διαδικασία που προτείνουμε καταργείται ο λόγος ύπαρξης της διαδικασίας 42.00. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ο τελευταίος λόγος ε, από τον εισηγητή, τον κύριο Λάγκεν. Θα είμαι σύντομος, θα ευχαριστήσω καταρχήν τους εμπειρογνώμονες. Έμαθα σήμερα ότι στην Τσεχία προφανώς υπάρχουν θετικές εμπειρίες που οδήγησαν δηλαδή σε συγκεκριμένες βελτιώσεις. Έμαθα επίσης ότι ένα βασικό πρόβλημα είναι η ελλειπής συνεργασία σήμερα, η ελλειπής αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας διασυνοριακά. Δεν ξέρουμε... Ε, ε, ε, ξέρουμε πόσο κρατάει αυτή η ιστορία, αλλά δεν θα μπορέσουμε στο δινικές να βελτιώσουμε το σύστημα αν δεν ασχοληθούμε με αυτό. Τώρα, ε, οι καταληκτικές παρατηρήσεις του εκπροσώπου του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν είναι ε, αυτό που λέει στο σημείο 89 ότι επιβεβαιώνονται οι επιφυλάξεις και ένας ε, συμμετέχον μόνο πρότεινε την αντιστροφή. Ναι, η Τσεχία βέβαια ήταν, το ΕΚΟΦΗΝ έκανε την ψηφοφορία και 10 ε, στήριξαν την πρόταση, την πρόταση όχι μόνο το πιλωτικό σχέδιο. 12 πέσχων οι άλλοι κατά. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας, της άτυπης ψηφοφορίας φέτος τον Ιούλιο στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Και αυτό που αναφέρεται εδώ, το αίτημα, δεν είναι το αποτέλεσμα που αναφέρεται στο κείμενο του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτό ήθελα να σας το πω. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα που συζητήθηκε, δηλαδή που είναι μεγαλύτερες οι δυνατότητες για απάτη. Δεν ε, ε, είναι στην εθνική αρμοδιότητα, γιατί φαίνεται ότι κάθε εθνικό κράτος ε, μπορεί να παρεμβαίνει ε, αυτόνομα και αυτό είναι ε, αυτό το σύστημα αν το εξετάσουμε και το ε, εγκρίνουμε θα μπορεί να ενισχύσει την δυνατότητα αντιμετώπιση σε εθνικό επίπεδο. Η ενιαία εφαρμογή θα ε, ε, ε, πρέπει να εξεταστεί. ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είχε πει κάτι, τον συνάντησα τον Απρίλιο, και είπε ότι η εισαγωγή των ηλεκτρονικών ταμείων σε ελληνικό εμπόριο, το ΦΠΑ, το αύξησε κατά 18%. Δηλαδή είναι στο χέρι των ε, εθνικών αρχών να καταπολεμήσουν την μαύρη ε, οικονομία και τις απάτες. Δεν ακούγεται καλά ο μιλητής που γυρίζει έτσι. Ε, θα πρέπει να, μέσα από αυτό το πνεύμα να δούμε και τις προτάσεις από τη Γερμανία, από την αστυνομία δίωξης του εγκλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω ότι στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με τους Σκιώδης θα προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση μιας καλής λύσης. Ευχαριστώ πολύ ε, και εγώ τους εμπειρογνώμονες για τις ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις τους σήμερα το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι της ημερήσιας διάταξης και προχωρούμε στο σημείο 7 ε, Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό έτος 2017, όλα τα τμήματα. Έχουμε και την εξέταση των τροπολογιών ε, και αύριο θα ψηφίσουμε. Δίνω άμεσα το λόγο στον κύριο Φέρμπερ, τον συντάκτη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Μετά τις θερινές διακοπές όλες οι επιτροπές καταπιάνονται με, το, τον προϋπολογισμό. Το προπολογισμό του 17 έχει μια ιδιαιτερότητα γιατί η Κομισιόν θεώρησε ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού θα έπρεπε να ε, προταθεί μετά τις 22 Ιουνίου. Έπρεπε κανονικά το Μάιο να γίνει αυτό. Διαπιστώσαμε όλοι ότι ήταν καλή και σωστή απόφαση γιατί ο Βρετανικός λαός... Ε, ε, ε, έλαβε τις αποφάσεις του. Ε, το, το είχαμε αναβάλει για να δούμε μήπως ο Βρετανικός λαός θα αποφάσιζε να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πάντως αυτό είναι το έγγραφο που χρησιμοποιούμε ως βάση για τις εργασίες μας τώρα που δεν υπευλήθη ο συνήθως στα πλαίσια των συνήθων προσθεσμιών. Ευχαριστώ πολύ του όσους ασχολήθηκαν με την έκθεση αυτή, διότι εργάστηκαν επικοδομητικά παρόλο το πρόβλημα με τα χρονοδιαγράμματα. Ε, μας δυσκόλεψε το γεγονός ότι έπρεπε να δουλέψουμε για μεγάλο διάστημα χωρίς νούμερα. Ήταν σημαντικό και πάνω στη βάση αυτών που κάναμε στα πλαίσια της απαλλαγής για τον περσινό προϋπολογισμό του 2015, ε, και είχα την τιμή να ήμουν ε, σκιώδης, ε, είχα αναλάβει το βάρος του σκιώδους, τους αδύναμους ώμους μου. Ε, πάντως ε, το, το ζητούμενο είναι να έχουμε ένα σχέδιο πολιτική συνεκτικό που θα αντικατοπτρίζει τις προθέσεις μας και τις πολιτικές μας. Έχουμε την ε, δημιουργία ικανοτήτων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ένα πιλωτικό πρόγραμμα και προπαρασκευαστικό σχέδιο. Η Κομισιόν τώρα έχει προτείνει νομική βάση που χρειαζόταν αλλά που πρέπει να εγκριθεί και σας ε, συστήνω στην Επιτροπή που είναι υπεύθυνη επί της ουσίας να δημιουργήσει αυτή τη βάση, αλλιώς δεν θα υπάρξουν χρήματα. Συμφωνήσαμε όμως ότι θα φροντίζαμε ώστε τα θεσμικά, ε, ε, ε, ώστε οι θεσμοί που θα ωφελούνταν να έχουν ίδιους σπόρους και να μην εξαρτώνται από τα ψίχουλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τρεις εποπτικές αρχές μας απασχόλησαν που ως έκον πρέπει να τις ελέγχομαι. Έκανα συζητήσεις από πριν και με τις τρεις και ε, με την ε, ΕΙΟΠΑ και... με τον αρμόδιο υπάλληλο για τον προϋπολογισμό στα πλαίσια των ε, αρχών των υποπτικών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την εποπτεία στον ασφαλιστικό τομέα. μόνο η ΕΣΜΑ που εποπτεύει τη αγορά αξιογράφων. Ε, εδώ μόνο δεν προβλέπεται αύξηση των ε, πόρων. Ε, για μένα ήταν σημαντικό να ξέρω και χαίρομαι που υπάρχει κομισιόν. Ήθελα να ξέρω τι θα εδικαιούνται οι αρχές αυτές σε σχέση με τον αριθμό των υπαλλήλων. Γιατί είχαμε κάποια σύνθετα συστήματα και απογοητεύτηκα γιατί τα τελευταία, τις τελευταίες 14 μέρες ε, δεν ε, βρέθηκε κανείς από την Κομισιόν να μου δώσει τα στοιχεία που έπρεπε. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Ε, Μία υποπτική αρχή ε, έχει την έδρα της σε χώρα που θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό νομίζω ότι ήδη από του χρόνου η ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα πρέπει να λάβει μέτρα για να φροντίσει ώστε να μην παραμείνει σε χώρα ε, που δεν θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, να, κάνουν, να λάβουν τα μέτρα που πρέπει για να προετοιμάσουν τις κινήσεις τους το, την επόμενη χρονιά. Τα τελευταία χρόνια επίσης ασχοληθήκαμε πολύ με το θέμα του φορολογικού δικαίου. Έχουμε ένα πρόγραμμα μέχρι το 2020. Ζητάμε η Κομισιόν να εξετάσει το θέμα στα πλαίσια του, των απορισμάτων τάξη 1 και 2, γιατί ήδη έχουμε ε, προεργασία στον τομέα της συνεργασίας στα φορολογικά θέματα. Έχουμε και το πρόγραμμα Φισκάλης που μπορούμε ίσως να το ε, διορθώσουμε λίγο, ούτω ώστε να ε, έχουμε και άλλες μορφές συνεργασίας. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να συμπεριληφθεί. Στον τομέα της φορολογικής διαφάνειας θα ήμουν ευτυχής αν είχαμε καταφέρει να έχουμε ένα προπαρασκευαστικό μέτρο. Η συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Τάξουντ ήταν λίγο απογοητευτική. Προτείνω να έχουμε συνέχιση μόνο ενός πιλωτικού μέτρου που θα συνεχιστεί. Θα ήθελα όμως μεγαλύτερη υποστήριξη από την Κομισιόν εδώ. Σε έφθετο χρόνο θα το συζητήσω και με τον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος είχε έρθει στην Επιτροπή και μας είχε πει πόσο θεωρεί σημαντική τη συνεργασία με την Επιτροπή μας μπορούμε να επιτελέσουμε πρόοδο στα φορολογικά. Ε, θα κάν, ε, κάναμε μια συνάντηση με τους συσκιώδεις όπου προσπάθησαν να επεξεργαστώ ε, συμβαστικές λύσεις με καλά αποτελέσματα και θέλω και να τους ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης για την επικοδομητική ατμόσφαιρα που επικράτησε, ώστε να μπορέσω αύριο να ε, υποβάλω ισορροπημένη πρόταση. Με μεγάλη υπευθυνότητα αντιμετωπίζουμε τα χρήματα των φορολογουμένων και στα πλαίσια του ψηφίσματός μας παρουσιάζουμε και κάποιες πολιτικές προτάσεις και ελπίζουμε ότι θα τις εγκρίνει το Κοινοβούλιο. Φυστώ την προσοχή σας σε αυτό. Ελπίζω μετά από δεκαετή παραμονή σε αυτή την Επιτροπή ότι είναι γνωστοί οι κανόνες του παιχνιδιού. Αυτά τα ολίγα από τη δική μου τη πλευρά. Ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε μία ισορροπημένη πρόταση που θα μας βοηθήσει στα πλαίσια της διαδικασίας προϋπολογισμού του 2017. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Τώρα με τη σειρά Η Περβάνος Περέζε για τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες αντικαθιστά του Σκιώδη. Ο κ. Κοτσολίνο ζητά συγγνώμη γιατί χρειάστηκε να επιστρέψει στην Ιταλία εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων. Μου ανέθεσε να σας ευχαριστήσω θερμά ε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους άλλους και εισηγητές για την συνεργασία, για όλη τη δουλειά τους σε αυτό το ζήτημα. Ε, επιθυμεί να κάνω τέσσερα σχόλια, πέντε σχόλια συγγνώμη. Πρώτον, ε, θέλουμε να υπογραμμίσουμε το θέμα της, των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Για την δική μας πολιτική ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί αυτό το κεφάλαιο. Ε, το κονδύλι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ε, για να εργαστούμε υπέρ των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Της ανάπτυξης της καινοτομίας, της, ε, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Όλα αυτά είναι οι προτεραιότητες μας και ο στόχος πρέπει να είναι το ύψος των επενδύσεων να φτάσει ξανά στα επίπεδα που βρισκόταν πριν την κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ίδιο πνεύμα πρέπει να στηρίξουμε την δυνατότητα παρέμβασης και τις δραστηριότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω δράσεων που θα ενθαρρύνουν και θα βελτιώνουν την ανάπτυξή τους και την ανταγωνιστικότητά τους. Δεύτερο σημείο, η ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της στήριξης των οργανισμών που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Ε, εμείς ε, ε, δεχόμαστε τις επισκέψεις και τις παρενοχλήσεις διαφόρων λόμπι που έχουν πολύ ισχυρά μέσα. Πρέπει να στηριχθούν και οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που έχουν λιγότερα μέσα, διότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των καταναλωτών, στην ε, και στην, στο σχεδιασμό ε, νομοθεσίας, ε, ισόρροπης νομοθεσίας. Μόνο αν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα μπορούν να κάνουν το έργο τους και να πετύχουν τους στόχους τους. Τρίτον, θα πρέπει ε, η, να όλες οι υπηρεσίες της ε, Κομισιόν να έχουν επαρκή μέσα και προσωπικό. Θα πρέπει να βρεθεί ένας, μια ισορροπία. Τέταρτον, ο κ. Κοζολίνο και η Σοσιαλιστική Ομάδα επιθυμούν διακαώς να καλέσουν τον εισηγητή να ξαναδεί την παράγραφο 5 που αμφισβητεί τις δραστηριότητες των υπηρεσιών ε, της Ευρωπαϊκής ε, ε, θα θέλαμε να διαγραφεί αυτή η παράγραφος. Τέλος, ο κ. Κοζολίνο υποβάλλει τη, μια τροπολογία σε ό,τι αφορά την εύση. Θα θέλαμε να στηριχθεί ε, προκειμένου να δώσουμε όθηση στις επενδύσεις ε, και στην ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βλέπω άλλους σκιώδεις. Δεν βλέπω εκπροσώπους του ECR. Α, η φιλελεύθερη. Αντί για τον κύριο Τόρβαλ, κυρία Φαν Χουμπερνχόλζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Ο κύριος Τόρβαλτς μου ζήτησε πρώτα-πρώτα ε, τον συγχωρείτε που δεν ήρθα εδώ γιατί είχε κάποια υποχρέωση δυστυχώ. Αλλά μου είπε να σα διαβάσω το εξή μήνυμα. Είναι θετικό ότι συμφωνεί με όλε τι συμβαστικέ τροπολογίε. Αυτό και τίποτε άλλο. Καλά τα νέα σα Για την ΚΟΕ, ο κύριος Κράσπο. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται το Brexit να γίνει ούτως ώστε να καταλάβουμε ότι βρίσκεται σε βαθιά κρίση η Ευρώπη. Έχει αντιμετωπίσει χιλιάδες προσφύγων, μεγάλη ανεργία στο Νότο και τροπεζικό σύστημα το οποίο έχει χτυπηθεί από την κρίση όπως είδαμε από τα τελευταία stress tests. Όλα αυτά τα προβλήματα που δείχνουν ότι χρειάζεται δράση συντονισμένη η Ευρώπη και χρειάζονται οι πόροι για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Να μην κατησχίσει ε, το ιδιωτικό συμφέρον και μια κοντόφθαμη λογική. Όμως, ε, τι είχαμε εδώ πέρα, είχαμε 2% περικοπή ε, στους πόρους που επιβλήθη δύο φορές έτσι λέει το σχέδιο προϋπολογισμού. Όμως το θέμα ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το ευρωπαϊκό εξάμεινο, τι γίνεται με το πρόγραμμα προσαρμογής. Αυτό μας οδηγεί σε ανεργία, σε στασιμότητα και όλα αυτά είναι αφόρητα. Επομένως, έχουμε αυτό το πολιετές δημιουργικό πλαίσιο. Αυτό είναι πάρα πολύ περιοριστικό και μας ε, οδηγεί σε κατάσταση πολύ διαφορετική από ό,τι προβλέπει το πλάνο Juncker για τους ιδίους πόρους. Άρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα βγούμε από την κρίση, αλλά σίγουρα όχι με αυτόν τον υπολογισμό που μας ε, στέλνει στην αντίθετη κατεύθυνση. Επομένως χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Ευχαριστώ συνάδελφε Κρέσπο για τους πρασίνους. Τώρα, ε, ευχαριστώ πολύ Ελπίζω να περάσατε ωραία το καλοκαίρι σας. Τώρα, να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή για τη συνεργασία. Υποστηρίζουμε όλες τις συμβιβαστικέ προτάσεις όσες έχουν τώρα. Ξανατονίζω ότι ο ρόλος της νομοδότησης δεν είναι να έχουμε γενική συζήτηση για τον προπολογισμό. Μπορεί να γίνει και αυτό, γιατί υπάρχουν πολλές απόψεις μας που μπορούσαμε να μοιραστούμε εμείς οι πράσινοι, αλλά δεν είναι δουλειά μας αυτή. Τέλος, να ζητήσω από όλες τις ομάδες, γιατί υπάρχει ε, μία αναφορά στο προπολογισμό της Eurostat. Θέλουμε να ε, παληθεί η αναφορά στην κοινωνική οικονομία και την μη ε, ε, συμμόρφωση προς το ε, στατιστικό πρόγραμμα που από κοινού συμφωνήθηκε στη Eurostat. Νομίζω ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Καλό λοιπόν όλες τις ομάδες Α, η πρόταση ήταν για ε, απάλληψη, αλλά ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να παραμείνει αυτή η διατύπωση, γιατί είναι σημαντική για τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ Κομισιών και Eurostat για να πληρούνται οι όροι και οι αιτιολογήσεις. Όχι απάλληψη λοιπόν της κοινωνικής οικονομίας. Κατά τα άλλα συμφωνώ και θα υποστηρίξουμε την έκθεση. Ευχαριστώ συνάδελφε Γκίγκολτ. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Η, σκιο... Α, η κυρία Κάπαλγε, την Ευχαριστώ. Και εγώ νομίζω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα αύριο. Είναι ισορροπημένη η ε, ε, πρόταση, το κείμενο. Έχουν τεθεί σωστά οι προτεραιότητες σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις προτεραιότητές τους, αύξηση της επενδυτιστικής δραστηριότητας. Ε, υπάρχει ακόμα ε, ένα κοινό 400 δις ευρώ. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα με βάση τις ε, συστάσεις αναχώρα είναι σημαντικό να εφαρμοστούν όπως και μια ισορροπημένη πολιτική δημοσιονομική. Αυτά ελήφθησαν υπόψη. Τώρα για τις ε, δυνατότητες κοινωνίας των πολιτών είναι σημαντικό εδώ ο βαθμός χρηματοδότησης ε, να αλλάξει. Εδώ έχουμε 50% δημόσιο, στο δημόσιο. Χρειάζεται μεγαλύτερη ε, προσπάθεια για τις ε, τρεις αρχές, εποπτικές αρχές. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να περιορίζονται στις δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί και ενδεχομένως θα πρέπει να φύγει η ΕΜΠΑ από το Λονδίνο. Πρέπει να ε, αρχίσουν να λαμβάνονται μέτρα από τώρα. Αύριο, κατά τα άλλα, νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει να λάβει το λόγο τώρα. Όχι. Άλλες παρεμβάσεις δεν έχω. Οπότε δίνω το λόγο στον εισηγητή για να κλείσει το θέμα. Ευχαριστώ. Ε, να πάρω στοιχεία από την Κομισιόν που τα περιμένω εδώ και εβδομάδες. Δεν τα έλαβα. Ε, λίγες παρατηρήσεις θα κάνω. Συνάδελφε Κρέσπο, εμείς... Ε, Είμαστε μια επιτροπή γνωμοδοτική. Αυτό το κοινοβούλιο ε, δέχτηκε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, η ομάδα σας όχι. Εντάξει, αυτό δεν πειράζει, αλλά πρέπει να σεβαστείτε το γεγονός ότι δεχτήκαμε το δημοσιονομικό πλαίσιο, στα πλαίσια του κινούμεθα και γι' αυτό ήταν δύσκολο να βρω συμβαστικέ λύσει με την ομάδα σα. Γιατί σήμερα δεν μιλάμε για την αλλαγή του δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά για τις γραμμές του προϋπολογισμού που είναι αρμοδιότητα δική μας. Στα πλαίσια της γενικής συζήτησης, την επόμενη εβδομάδα μετά τη δήλωση Γιούγκαρ ή στα πλαίσια της ενδιάμεσης αξιολόγηση του δημοσιονομικού πλαισίου που ε, ε, θα γίνει, μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Όχι όμως τώρα. Για την παράγραφο 5 θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ ΕΛΚ και Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Αύριο θα ψηφίσουμε και θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Ε, όλα πρέπει να τα εξετάζουμε με την προοπτική μιας συμβιβαστικής λύσης. Καμιά φορά βέβαια χρειάζεται να λύσει το θέμα και η ψηφοφορία, όπου η πλειοψηφία θα αποφασίσει. Για τον συνάδελφο Γκίγκολτ μια παρατήρηση. Εδώ το θέμα είναι με ποια κριτήρια μπορεί να απελευθερωθεί ένα αποθεματικό. Εγώ είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ ε, για το αποθεματικό, αλλά θα προσκρούσουμε σε αντιρρήσεις. Θυμάμαι στην Επιτροπή Προϋπολογισμών που είχαμε κάποια μικρά ποσά στο αποθεματικό και Βλέπαμε ότι παρόλα αυτά το Συμβούλιο ε, έκανε στροφή 180 μοιρών σε σχέση με τα συμφωνημένα γιατί τον ενδιέφερε πολύ η μία γραμμή του προϋπολογισμού. Εγώ εκτιμώ, αυτό το αποφασίζει η πλειοψηφία, ότι η αυτή η προϋπόθεση ξεπερνάει αυτά που ε, συμπεριλαμβάνονται στην συνένεση που βρήκαμε. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό θα το αποφασίσει αύριο η πλειοψηφία. σωστό είναι για να καταλήξουμε κάπου. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και το καλό κλίμα. Γιατί ήταν λίγο αστεία η διαδικασία για τον προπολογισμό, αφού δεν είχαμε στοιχεία, αριθμητικά στοιχεία. Όμως, παρόλα αυτά, ε, θεωρώ ότι αύριο θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε μια καλή συμβιβαστική λύση η οποία θα έχει θετικό αντίκτυπο, ε, όπως ελπίζω, και στην Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τώρα πάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Ε, πάλι ε, εξέταση τροπολογιών, πράσινη βίβλου για τις λιανικές χρηματοστατικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 28 Ιουνίου ήταν η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Ο εισηγητής ε, Όλε Λούντβιξον έχει το λόγο. Όλε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως τα γνωρίζετε, σίγουρα, βέβαια γυρίσαμε από τις διακοπές και τώρα ασχολούμαι με αυτή την πράσινη βίβλο για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που αφορούν και τις ΜΜΕ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι γιατί οι τροπολογία ήταν πολύ ενδιαφέρουσες όλες όσες έχετε υποβάλει. Είναι ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό, επομένως ξεκινάμε με το δεξί την προβληματική και έχουμε διάφορες ε, ιδέες που πέσανε εδώ που είναι πάρα πολύ θετικές. Πιστεύω θα έχουμε αγαστή συνεργασία και θα έχουμε κάποιες λογικές συμβαστικές τροπολογίες και ότι όλες οι περιοχές του Κοινοβουλίου θα μας βοηθήσουν. Εγώ θέλω τώρα να σας τονίσω ότι η μεταξύ μας συνεργασία πρόκειται να συνεχιστεί. Θα έχει εντατικό χαρακτήρα, γιατί έχουμε πάρα πολύ ποιοτικέ τροπολογίε και ελπίζω ότι η συζήτηση την οποία θα κάνουμε πρόκειται να καλύψει όσο γίνεται περισσότερε από αυτέ τι τροπολογίε και έτσι να έχουμε όσο γίνεται πιο ευρεία ε, συμφωνία. Ε, θα πρέπει να επικρατήσει πνεύμα θετικό, να καταλήξουμε σε αξιόλογες συμβαστικές τροπολογίες. Θα πρέπει και η συζήτηση να έχει επικοδομητικό χαρακτήρα, αλλά επίσης θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και να έχουμε πρακτικό πνεύμα στις τροπολογίες μας για να μπορέσουμε να πάρουμε ψήφους από όλες τις πέργες. Υπάρχουν εδώ πολύ σημαντικά προβλήματα που πρέπει να επιληθούν Επίσης ε, ε, υπάρχουν εδώ πέρα αντίθετες απόψεις, δεν μπορούμε να τις ε, συγκεράσουμε όλες παρόλα αυτά. Εγώ ελπίζω ότι τελικά θα βρούμε τη μέση οδό. Στην Επιτροπή μας θα διαμορφώσουμε τελικά μία γνωμοδότηση που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ, θα αποτελεί μία προσθεμένη αξία. Το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτει πάρα πολλούς από τους εμπλεκομένους, πάρα πολλούς τομείς που διέπονται από διαφορετικές συνθήκες γιατί αναπτύσσονται σε διαφορετικές χώρες. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι η διασυνορική συνεργασία γίνεται ή μπορεί να γίνει σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά αυτή την υπόθεση πριν νομοθετήσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ανάλυση και συλλογή ε, αξιοπίστων στοιχείων και δεδομένων και έτσι να έχουμε μια στερεή βάση. Έχω πέντε θέματα να σας αναπτύξω. Πρώτα-πρώτα έχουμε μια σειρά τροπολογιών που αφορούν κάποια θέματα που είναι στενά εθνικού χαρακτήρα. Δεν θέλουμε να εντείνουμε τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά. Βέβαια έτσι θα έχει ο καταναλωτής καλύτερη τιμή, καλύτερα προϊόντα. Όμως έχουμε κάποιες τροπολογίες που κάποιες φορές είναι αντιφατικές, άρα δεν θα πρέπει να κολλήσουμε σε αυτά τα εθνικά ζητήματα, σε εθνικές ιδιομορφίες. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Επιτροπή να δημιουργήσει περισσότερο ανταγωνισμό καλύτερη εσωτερική αγορά. Να μην υπάρχει προστατευτισμός για κάποιους ε, συνεργασόμενους σε εθνικό επίπεδο. Άρα θα πρέπει να μην δοθεί προτεραιότητα σε κανέναν παρά μόνο στον καταναλωτή. Προέχουν τα συμφέροντα του καταναλωτή. Αυτές οι τροπολογίες είναι οι σωστές. Άρα θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε αυτές τις τροπολογίες. Γιατί όταν έχουμε διανομής και προμηθευτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βρίσκεται πολλές φορές τριμωγμένος ο καταναλωτής. Αυτό αφορά και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Άρα έτσι θα πρέπει να αναβαθμίσουμε την προστασία του καταναλωτή. Και όσο πιο πολύ προστατεύσουμε τον καταναλωτή, τόσο καλύτερα θα λειτουργεί η ενιαία αγορά. Έτσι θα έχουμε πιο υγιή ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά. Δεν θα έχουμε περιθωριοποιήσεις οικονομικές. Λέμε επίσης για τις προκλήσεις ε, τις ψηφιακές. Να μην τις υποτιμούμε. Πολλοί πρέπει να εκπαιδευτούν, να μάθουν καλύτερα για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή τους. Οι πιο ηλικιωμένοι δυσκολεύονται, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις νέες ευκαιρίες που υπάρχουν. Να δούμε πώς με τις καινοτομίες θα βελτιώσουν την εσωτερική αγορά και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, Να μην υπερεκτιμούμε βέβαια και τις ψηφιακές δυνατότητες. Θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν ε, προϊόντα τα οποία να είναι φιλικά στην χρήση τους. Η χρηματοπιστωτική τεχνολογία, fintech, μπορεί να αξιοποιηθεί από την ενιαία αγορά και η παραδοσιακή συναλλασσόμενη μπορούν να βοηθήσουν τον καταναλωτή, αλλά και να δημιουργήσουν θέσει απασχόληση για την Ευρώπη. Βέβαια, και υπάρχει η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι εμπλεκόμενοι από την παγκόσμια αγορά εκτός Ευρώπης. Πάντως η εσωτερική αγορά θα πρέπει να ωφελεί τους καταναλωτές. Και εδώ υπάρχουν οι δυνατότητες ούτως ώστε να υπάρχει διεθνοποίηση του κάποιων ε, τομέων. Άλλο γίνεται αυτό, άλλο δεν γίνεται. Θα πρέπει τέλο πάντων εμεί να εξισορροπήσουμε όλα αυτά τα επιμέρου ζητήματα. Προσφέρονται εδώ πολλέ ευκαιρίες αλλά υπάρχουν και οι δυσκολίε σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να γενικολογούμε ούτε να υπεραπλουστεύουμε ούτε μπορούμε με την εναρμόνιση να υπονομεύουμε το φορολογικό σύστημα των κρατών μελών ή χειρότερα να διακυβεύουμε την χρηματοοικονομική σταθερότητα των κρατών μελών. Άρα θα πρέπει να δούμε και κάποιες λεπτομέρειες, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα χαμηλά επιτόκια που είναι γεγονός της σημερινής συγκυρία. Ε, αυτό σίγουρα θα επιδράσει στην βιωσιμότητα της αγοράς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές τροπολογίες κολλάνε σε πολύ συγκεκριμένα, πολύ περιορισμένα θέματα. Θα πρέπει να υπάρχει ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων την, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να είναι στεγανή, προσεκτική. Θα πρέπει επίσης και εμείς να προσπαθήσουμε ούτως ώστε να έχουμε ένα κείμενο που θα βοηθά και θα βελτιώνει την κατάσταση. Ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες που θα συνεργαστούμε όλα να είναι επικοδομητικά. Πολύ σημαντικό επίσης και το κείμενο, η πράσινη βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση ως Κοινοβούλιο να βοηθήσουμε να έχουμε δημιουργική στάση και να βελτιώσουμε τα πράγματα και να μπορέσουμε να συντάξουμε έκθεση που να την υποστηρίξει όλο το Κοινοβούλιο. Να μπορέσουμε να βρούμε κάτι που να είναι προστιθέμενη αξία, να ωφελεί τους καταναλωτές να πάμε προς σωστή κατεύθυνση με τροπολογίε που θα τι υποστηρίζουν όλοι και έτσι να ωφεληθούν οι καταναλωτέ Από αυτή την οπτική αγωνία βλέπουμε τα πράγματα. Να είναι φθηνότερε οι χρηματοπιστωτικέ εν λόγω υπηρεσίε. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή, Όλε. Περνάει ο χρόνο, οπότε να περιορίσουμε στα τρία λεπτά το χρόνο των αναπληρωτών. Ε, ο κύριος Μπάλτς πρώτος. Όχι, όχι, δεν ε, τον αντικαθιστώ τον κύριο Μπάλτσα, εδώ είναι. Είμαι όμως και ο συζητητής. Να είναι εδώ είμαι, εδώ κάθομαι. ο κύριος Καντέκ. Α, δεν σας είδα, δεν σας συμπαθάτε με. Δεν με βλέπετε συχνά, είναι αλήθεια εδώ στην ΕΚΟΝ. Γιατί είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Αλίας, ε, γι' αυτό και δεν έρχομαι εδώ συχνά. Όμως παρακολουθώ προσεκτικά τις εργασίες της Επιτροπής μας. Οπότε είμαι για το Λαϊκό Κόμμα ως κοιόδης εισηγητής. Θεωρώ ότι είναι δύσκολη υπόθεση ε, το θέμα που ρυθμίζει η Πράσινη Βίβλος και βέβαια να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Λούντβιξον ε, για τη δουλειά του. Πρώτα πρώτα. Κοιτάξτε έχουμε ένα σωρό εμπόδια για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική αγορά λιανικών χρηματοπιστών υπηρεσιών. Είναι και πολιτιστική φύσεω και χρηματοπιστωτική αυτέ οι δυσκολίε. Επίση, δεν θα πρέπει να βιαστούμε. Γιατί έχουμε πάρα πολλά νομοθετήματα που βρίσκονται στη φάση της μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο. Θα πρέπει επομένως να μην βιαστούμε, να αναλύσουμε ποια είναι τα πάγια εμπόδια για αυτές τις διασυνοριακές συναλλαγές. Επίσης θα είναι αντιπαραγωγική η ομοιογενής αντιμετώπιση γιατί έχουμε μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα και στους εμπλεκομένους. Μια ευρωπαϊκή ε, αγορά για λιανικές υπηρεσίες τέτοιες ωφελεί τους καταναλωτές αλλά και τους επενδυτές αλλά και τις επιχειρήσεις. Το είπε ο συνάδελφος, έχουμε μια σειρά από τοπολογίε που ζητούν να μην ε, ξεχάσουμε στο νομοθέτημα αυτό τους κανόντες θα πρέπει να μπορούν να έχουν φιλικές υπηρεσίες, εύκολη προσβασιμότητα και μη και ο καταναλωτής για αυτές τις υπηρεσίες και αυτό θα πρέπει επίσης τη, τη, τη, την χρηματοπιστωτική κουλτούρα να βελτιώσουμε και για το ΕΛΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό μια τέτοια αγορά να βελτιώσει την προσβασιμότητα για τις ΜΜΕ ε, και διασυνοριακά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη και να υπάρχει ε, ανταγωνισμός με θεμητές ε, συνθήκες και βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες που πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα η ψηφιοποίηση επίσης ε, είναι μια επανάσταση πολύ σημαντική για τον τομέα αυτών των υπηρεσιών. Θα πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες καινοτομίας που προσφέρονται. Είπαμε ότι χρειάζεται ευελιξία στην νομοθεσία και θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της καινοτομία. Είπαμε για τις συναλλαγές τις διασυνοριακές, αλλά θα πρέπει να έχουν περισσότερη, καλύτερη ταυτοποίηση και να μην φύγεται το θέμα της ασφάλειας των συναλλαγών. Άρα όσον αφορά τον καταναλωτή, πολλοί λένε ότι θα πρέπει οι λιανικές αυτές υπηρεσίες να μην είναι περίπλοκες. Έχουν δίκιο. Συμφωνώ θα πρέπει να προχωρήσουμε όπου γίνεται ή που δεν γίνεται πάντοτε σε απλούστευση σύγκριση. Να μετράτε η ποιότητα των υπηρεσιών, να μην έχουμε μοναδικό κριτήριο τη τιμή των υπηρεσιών. Προσοχή. Θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν ούτως ώστε να καταλήξουμε σε κάποιο είδους διακρίση διακρίσεις επί τη βάση του τόπου κατοικίας. Ε, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί γεωγραφικοί ε, που αφορούν κάποια κρατημέλια. Από αυτό δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Δεν θα πρέπει επίσης να είναι εμπόδιο για το να καταλάβει το προϊόν ο καταναλωτής η ποσότητα των πληροφοριών. Θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο, λένε σε πολλές τροπολογίες, περισσότερη εμπλοκή των εποπτικών αρχών. Τώρα αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τις διασυνορικές συναλλαγές. Όλα αυτά τα στοιχεία να ληφθούν υπόψη και θα συνεργαστούμε με τους σκιώδες ηγητές και τον εισηγητή για άλλη μια φορά να τον ε, ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φόξ, Άχλη Φόξ η Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λούτινγκσον για το προσχέδιο έκθεσης ε, και τους συναδέλφους για τις τροπολογίες τους. Η δική μου, ο δικός μου στόχος είναι ε, μια, ένα πλαίσιο ε, ανταγωνιστικό και ανεξάρτητο τεχνολογίας. Αυτό θα επέτρεπε την ανάπτυξη τόσο των μικροψηφίων επιχειρήσεων όσο και των νεοφύων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ε, σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που ήδη υπάρχουν και είναι επιτυχημένες θα προωθηθούν. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, το, οι προτεραιότητες, το πλαίσιο που έχει οριστεί ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τις μικρές και τις νέες επιχειρήσεις. Ε, οι μελλοντικές, το μελλοντικό ρυθμιστικό πλαίσιο ε, θα πρέπει να είναι ευέλικτο και να μην εμποδίζει την τεχνολογική ανάπτυξη. Στηρίζω την, τον αποκλεισμό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από το οργανισμό Geoblocking. οι τροπολογίες που ζητούν ενιαία αγορά για τα στεγαστικά δάνεια με προβληματίζουν. Χρειάζεται να δούμε πρώτα τι γίνεται με την, τον αντίκτυπο της ε, οδηγίας για τα στεγαστικά δάνεια. Πολύ λίγοι άλλωστε καταναλωτέ θέλουν στεγαστικό δάνειο σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο θα πληρώνουν. Επίση, ε, δεν θα, μάλλον επιφυλακτικό έναντι ε, τη ε, έναντι νομοθέτησης για πρόστα προϊόντα. Ε, τα... Επίσης είναι πολύ σημαντική η πληροφορία που θα δίδεται. Η, η τροπολογία 97 αναφέρεται στα προσπέκτους. Ε, είναι σημαντικό ότι τα KIDS και η τα προσπέκτους είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ε, ορισμένες, ε, ορισμένα προϊόντα δεν εμπίπτουν στην πρίψη αλλά χρειάζονται προσπέκτους. Ε, αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Στις ε, μελλοντικές συνεδριάσεις των συσχεωδών εισηγητών θα είμαι πρόθυμο να συζητήσω αυτά τα θέματα με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Η κυρία Ινβέλτ για, τους, ε, για την φιλελεύθερους. Ε, ευχαριστώ τον εισηγητή. Θα είμαι σύντομη. Αν ε, ξεκινούσαμε από το μηδέν, ε, θα αντιλαμβανόμουν τους ε, ενδιασμούς. Να σας δώσω κάποια στοιχεία όμως. Το πρώτο τρίμηνο του 2016 η χρηματοδότηση στην Ευρώπη είναι 350 εκατομμύρια δολάρια, ενώ είναι 2 δις στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια στην Κίνα για την χρηματοοικονομική τεχνολογία. Ε, οπότε καταλαβαίνω πολύ τι κοινωνικέ, τι πολιτικέ διαφορέ κλπ. Αλλά οι ανταγωνιστέ μα δεν ενδιαφέρονται για όλα αυτά. Οπότε ε, καταλαβαίνω τον εισηγητή και τον ενθαρρύνω να ακολουθήσει μια γενναία προσέγγιση, μια τολμηρή προσέγγιση γιατί χρειαζόμαστε την εσωτερική αγορά. Συμφωνώ με ορισμένα όπως είπε ο κ. Φόξ, αλλά διαφωνώ με το εξή. Ε, οι πολίτες μας ε, μπορεί να έχουν κάποιους συναισθηματικούς λόγους να είναι συνδεδεμένοι με ένα νόμισμα συγκεκριμένο, αλλά αν το στεγαστικό τους είναι 30% φθηνότερο με ένα άλλο νόμισμα, πιστεύω θα το σκεφτούν και θα δημιουργηθεί ενδιαφέρον. Δεν καταλαβαίνω γιατί να δημιουργούμε φραγμούς ρυθμιστικούς ή άλλους που ε, δεν εξυπηρετούν τους πολίτες και εξυπηρετούν μόνο τους πολιτικούς. Τα πράγματα κινούνται ταχύτατα στον κόσμο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας. Οπότε εμεί δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Ε, δεν έχουμε δικαίωμα να φοβόμαστε το μέλλον. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και να καταργήσουμε τα, τους περιττούς φραγμούς. Οπότε ενθαρρύνω τον συγητή να ακολουθήσει μια τολμηρή προσέγγιση. Ε, κύριε Ματίας, για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ τον συγητή. Συμφωνώ εν μέρη με, τον, με τα όσα είπε. Ε, με ανησυχούν όμως κάποιες τροπολογίες. Θα ήθελα να τις μοιραστώ τις ανησυχίες μου μαζί σας. Ε, έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από την αρχή της κρίσης και η εντύπωσή μου είναι ότι ακόμα δεν έχουμε διδαχθεί όλα όσα έπρεπε. Είναι τρομακτικό που συζητούμε αυτή τη στιγμή την χρηματοπιστωτική, τις ρυθμίσεις που θα βασίζονται στο ότι ε, η καινοτομία εκεί είναι κάποιες ιδέες μόνο. Ε, δεύτερον, ότι ε, οι νέες τεχνολογίες θα κάνουν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πιο διαφανείς. Εγώ τα βλέπω διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας και πάνω απ' όλα οι καταναλωτές θα ε, ήταν σε καλύτερη θέση αν η Λιανική Τραπεζική ήταν πιο συντηρητική. Η συντηρητική πλειοψηφία των καταναλωτών, αυτό που χρειάζονται είναι βασικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Και ε, ο, το καθήκον ε, των εθνιστικών αρχών είναι, των εποπτικών αρχών, είναι ε, οι καταναλωτές να μην βομβαρδίζονται από προϊόντα τα οποία δεν καταλαβαίνουν και είναι επικίνδυνα. Το πλαίσιο της κρίσης δεν ε, βλέπουμε ότι η τραπεζική κινείται σε φρενήρες ρυθμούς. Ο νομοθέτης όμως θα έπρεπε να την κάνει όσο πιο βαρετή γίνεται. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Ε, η, η ιδέα ότι χρηματοπιστωτική τεχνολογία θα επιτρέψει στους καταναλωτές να καταλάβουν αυτά τα περίπλοκα προϊόντα και να τα αναλύσουν είναι ε, Δεν είναι δυνατόν αυτά τα προϊόντα να πολλούνται στη λιανική τραπεζική. Ε, έχουμε δύο προτεραιότητες. Ε, οι εμπορικές τράπεζες δεν θα πρέπει να διακινούν ε, τέτοιου είδους ε, περίπλοκα προϊόντα θα πρέπει να μπορούν να διακινούν μόνο ένα περιορισμένο αριθμό προϊόντων ε, που καλύπτουν το 99% των αναγκών των καταναλωτών. Με αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες θα γίνουν πιο ασφαλείς, θα μειωθούν οι απάτες και θα ε, προωθεί ο ανταγωνισμός. Δεύτερον, δεύτερη προτεραιότητα, ε, η, η προσπάθεια ε, να κατηγορηθούν έμεσα οι εργαζόμενες τράπεζες για τις ανευθυνότητες που έχουν πράξει οι τράπεζες είναι λανθασμένοι και καταδικασμένοι. Ασφαλώς και θα πρέπει να διωχθούν ε, οι απατεώνες αλλά ε, όταν οι τράπεζες προσπαθούν να ταΐσουν στους ε, πελάτες τους προϊόντα τα οποία οι προελάτες αυτοί δεν καταλαβαίνουν, την ευθύνη την έχουν οι τράπεζες. Τρίτον, το γεγονό, η ιδέα ότι οι νέε τεχνολογίε θα κάνουν το τραπεζικό τομέα πιο διαφανή, ε, να πω το εξή. Η ταχύτητα με την οποία γίνονται οι, οι, συναλλαγές ε, καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο του τραπεζικού τομέα ακόμα και με τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών. Τελειώνω λέγοντας ότι οφείλουμε στους καταναλωτές να, απλοποιη... την... στους να απλοποιήσουμε και να καταστήσουμε πιο διαφανή ε, την τραπεζική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Ζήμων. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το καλό σχέδιο και την εισαγωγή που μας έκανε. Βλέποντας τις τροπολογίες, παρατηρώ πολλά κοινά στη βασική προσέγγιση πολλών τροπολογιών. Υπάρχει θετική στάση υπέρ της διασυνοριακής συνεργασίας, ε, της μεγαλύτερης, οι διαφορές δεν είναι μεγάλες, όπως έδειξαν ίσω κάποιες παρεμβάσεις εδώ. Θέλω να σχολιάσω κάποιες, κάποια επίμαχα θέματα. Άκουσα τη Μαρίζα αλλά διαφωνώ με την ανάλυση της. Ουσιαστικά, η 51 της Γκουε και αυτά που άκουσα τώρα λένε ότι αν υπάρχει λιγότερη διασυνοριακή δραστηριότητα θα είναι καλύτερο για τους καταναλωτές. Αυτό είναι λάθος νομίζω. Μου φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη συγκρισιμότητας προϊόντων, έλλειψη ανταγωνισμού και έτσι ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι υπερμεγέθης και πληρώνουμε υπερβολικά ως επενδυτές για το σύστημα διαμεσολάβησης. Έτσι, η μεγαλύτερη τυποποίηση και ανταγωνισμός μπορούν να βοηθήσουν για να μειωθούν οι τιμές και να συρρυκνωθεί ο υπερμεγέθης χρηματοπιστωτικός τομέας. Η προσέγγιση σας ουσιαστικά βοηθάει μόνο αυτούς που πληρώνουν σε βάρος των επενδυτών. Παρόμοια λάθος λύση, θεωρώ, είναι και οι τροπολογίες που θέλουν να περιορίσουν την ανάληψη κινδύνων από απλούς πολίτες. Υπάρχει από τους συναδέλφους από την EFTP, αλλά υπάρχει και από τον Γιάκοπ Φον Βάιτσεκερ μια τροπολογία παρόμοια και θέλω να το συζητήσω μαζί του. Και οι απλοί άνθρωποι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ανάληψη κινδύνου. Για παράδειγμα, αν είναι ας πούμε σε μια συνεταιριστική τράπεζα. Δηλαδή μετά τα ιταλικά προβλήματα πρέπει να απαγορεύσουμε στους απλούς πολίτες να γίνονται μέλη μιας ε, συνεταιριστικής τράπεζας και να ε, συστήνουν τράπεζα συλλογικά. Όχι. Αυτό που πρέπει να περιοριστεί και περιορίζεται ήδη από το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι να ε, συμβουλεύσετε να μην ρισκάρουν υπερβολικά μεγάλα εισοδήματα από αυτά που έχουν σε αυτούς τους τομείς. Δεν πρέπει να πάμε σε λάθος λύσεις όμως. Λίγες τροπολογίες ε, στηρίζουν περισσότερες βιώσιμες επενδύσεις και πράσινες επενδύσεις. Ε, γιατί υπάρχει το αυξανόμενο φαινόμενο fintech, χρηματοπιστωτική τεχνολογία δηλαδή, και θα πρέπει να το δούμε θετικά, γιατί είναι μια ευκαιρία για να ε, δημιουργηθεί πιο αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό τομέα που θα εξυπηρετεί καινοτόμε επιχειρήσει. Παράλληλα, θέλουμε υποστήριξη για τον ε, τομέα, τον διατηρήσιμο, βιώσιμο. Ε, αν θέλουμε... Ε, ένα λιανικό τομέα τυποποιημένο χρειάζεται και κοινή νομοθεσία και κοινή εποπτική κουλτούρα για την προστασία των επενδυτών. Και πολλές τροπολογίες εδώ κάνουν λάθος γιατί ζητούν περισσότερη διασυνοριακή δραστηριότητα αλλά σιωπούν ε, σε σχέση με την έλλειψη της προστασίας των επενδυτών. Αυτά πρέπει να συμβαδίζουν, γιατί αλλιώς ο κόσμος δεν θα εμπιστοευθεί ποτέ την διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Αλλά ελπίζω να βρούμε κοινό έδαφος. Ευχαριστώ πολύ. Μάρκο Να απαντήσω στον Σβέν γιατί αναφέρθηκε στην ε, Ιταλία. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση γιατί εκεί έχουμε πάρα πολλούς ε, που παρά την ΜΥΦΙΔ έχουν υποστεί απάντες και οι αρχές δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τους καταναλωτές. Εγώ διατηρώ κάποιε αμφιβολίες για όλες αυτές τις φιλοδοξίες που εξήγηλε η Σοφία Νετβέλτ. Αυτά είναι νεοφιλελευθερισμοί, γιατί τελικά ε, αυτά ε, τα, τα θέλουν οι κερδοσκόποι και όσοι, γιατί για τα μεγάλα συμφέροντα. Συμφωνώ με πολλούς από τους στόχους της πράσινης βίβλου, πρέσπιση του καταναλωτή κλπ. κλπ. Θέλουμε να υπάρχει ενή αγορά για αυτά τα προϊόντα, αλλά αυτό να μην είναι αντιπαραγωγικά γιατί θα πρέπει να προηγηθεί μία μεταρρύθμιση διαρθρωτική του τραπεζικού συστήματος. Να μην υπάρχει κερδοσκοπία, μην υπάρχει σκιώδης ε, οικονομία. Ε, τι γίνεται με τις εμπορικές τράπεζες, τι γίνεται με τα ταμιευτήρια. Προσοχή για την απορρίθμιση λοιπόν της ε, αγοράς κεφαλαίων. Προσοχή στην απορρίθμιση γιατί Τώρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η συμπλήρωση της ισχύουσης νομοθεσίας. Προσοχή στον αντίκτυπο. Να μην πληρώσουμε την ύφη επειδή δεν έχουμε φροντίσει κάτι. Ε, αυτό θέλω εγώ να τονίσω, αλλά βέβαια συμφωνούμε για την καινοτομία. Η καινοτομία θα πρέπει να μας προστατεύσει από, τους ρίσκους, από το ρίσκο κυρίως της απάτης προσοχή οι κίνδυνοι να εποπτευθούν και εκ των προτέρων να αποκλειστούν. Να έχουμε πιο αυστηρούς κανόνες για διαφάνεια ε, και για την ποιότητα των πληροφοριών που δίνουμε στον καταναλωτή για τα χρηματοπιστωτικά αυτά προϊόντα. Να ξέρει ο καταναλωτής τι ε, ρίσκο έχει κάθε του κίνηση. Ο μέσος άνθρωπος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για να μπορέσει να καταλάβει τι γίνεται. Θα πρέπει να του εξηγήσουμε. Πολλά προϊόντα είναι περίπλοκα από αυτά. Και η οικονομία είναι δύσκολη υπόθεση σήμερα. Πολλά από αυτά τα προϊόντα δεν εξυπηρετούν τον μικρό αποταμιευτή. Και ενεδρεύουν στην αγορά πολύ κίνδυνοι. Άρα να βρούμε έναν τρόπο ούτω ώστε να προστατεύσουμε αυτούς τους καταναλωτές. Να μπορέσουμε βέβαια να κάτσουμε στο τραπέζι και να τα συζητήσουμε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αλλά εμείς εμένουμε ότι πριν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση θα πρέπει να κάνουμε σοβαρές μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μην πάμε σε απελευθέρωση, ενώ ακόμα έχει πολλά παραθυράκια, πολλά κενά η νομοθεσία σχετική με τις τράπεζες. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάπελ έπρεπε κανονικά τώρα να λάβει το λόγο. Άλλος από την ΕΝΕΦ e δεν βλέπω να υπάρχει. Λοιπόν, ο εισηγητής για να συνοψίσει το θέμα αυτό. Όλε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Προσπάθησα να καταγράψω όλες τις απόψεις και γνώμες που ακούσαμε και θα προσπαθήσω να τις ε, σταθμίσω όπως πρέπει. Αυτή είναι πράσινη βίβλος, δεν είναι νομοθεσία. Η νομοθεσία θα έρθει αργότερα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε προσέγγιση προσανατολισμένη στο μέλλον. Μην κοιτάμε το παρελθόν, να δούμε το μέλλον, τι μπορούμε να φτιάξουμε. Η ιδέα κατ' εμέ είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες και καταναλωτές της ε, Ένωσης πρέπει να αποκομίσουν κάποια ωφέλη, κάποια πλεονεκτήματα μέσα από την αύξηση του ανταγωνισμού και να προωθήσουμε προϊόντα με τιμές προσιτές. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό προσπαθώ τουλάχιστον εγώ να κάνω στο έργο μου. Προσπαθώ να βρω λύσεις που μπορούν να στηρίξουν τους καταναλωτές αυτό είναι το πιο σημαντικό για τους καταναλωτές της Ευρώπης. Σε μια τέτοια διαδικασία δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα διαμιάς, θα πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Η συζήτηση είναι ότι, και θα την κάνουμε και αργότερα, ότι πρέπει να βρούμε τα σωστά βήματα. Τις επόμενες βδομάδες ε, περιμένω να στρωθούν τα πράγματα, να βρεθούν συμβιβαστικές. Είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να έχει μια φωνή και να, τύχει, να τύχουν προτάσεις ευρείας ε, υποστήριξης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλοι. 10-11 ε, Οκτωβρίου θα είναι η επόμενη επιτροπή και θα δούμε τι θα προκύψει. Σημείο 9 θέσπιση προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του ελέγχου από την περίοδο 2014-2020, ο εισηγητής ε, είναι ο Θείοντορ Δημητρού Στόλογιαν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. στηρίζω την πρόταση της Κομισιόν να, συνεχίσει, να συνεχιστεί η συγχρηματοδότηση ΕΦΡΑΓ την περίοδο 2017-2020 ούτως ώστε να ε, πραγματοποιηθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του προγράμματος Ένωσης και να υποστηριχθούν δραστηριότητες ε, για τη χρηματοοικονομική αναφορά και την ελεγκτική. Η ΕΦΡΑΓ είναι ιδιωτική κοκκύρος οργανισμός, ε, μη ε, ε, ε, δεν αποσκοπεί στο κέρδος, μη κερδοσκοπικός και χρησιμοποιεί διεθνή πρότυπα. Η διαδικασία έγκρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση του EFRS στηρίζεται στις, στην ομοδότηση της EFRAG. Ως εισηγητής πρέπει να σας θυμίσω τα εξής. Πρώτον, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης του EFRS και το PIOB, αποφασίσαμε για την ΕΦΡΑΓ το πρόγραμμα να καλύψει την περίοδο 2014-2016. Ε, ο σκοπός του ορίου αυτού ήταν να δούμε αν η ΕΦΡΑΓ θα εφάρμοζε τις ε, ε, συστάσεις της έκθεσης για την υποστήριξη και αύξηση της δραστηριότητας της ΕΦΡΑΓ. Δεύτερον, με βάση την αξιολόγηση της Κομισιόν και τη συζήτηση που είχαμε με την ΕΦΡΑΓ, μπορούμε να τονίσουμε ότι η ΕΦΡΑΓ εφήρμοσε τις περισσότερες συστάσεις της έκθεσης Μέσνερ. Αυτό που δεν μπόρεσε να εφαρμόσει η ΕΦΡΑΚ ήταν η σύσταση για την αλλαγή του χρηματοδοτικού μοντέλου της. Είχε συσταθεί ένα μοντέλο με βάση τη συνεισφορά των κρατών μελών ή τους, τους, δικαιούχους ε, της ΕΦΡΑΓ. Η εφαρμογή της σύστασης εξαρτάται όμως από τη βούληση των κρατών μελών. Η, η τροπολογία μου στην πρόταση της Κομισιόν υπενθυμίζει στην Κομισιόν ότι στην έκθεσή της ε, για την δραστηριότητα της ΕΦΡΑΓ και ΔΠΙΧ, και ΠΟΜΠ θα πρέπει να υποβάλει έκθεση και για τις συστάσεις σχετικά με τη δραστηριότητα της ΕΦΡΑΓ όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το σχετικό ψήφισμα από 7 Ιουνίου του 2016 για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, την ε, αξιολόγηση και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος ΕΦΡΑΓ ε, και της ε, PIOB. Ευχαριστώ. Υπερβάνους Περέσια του τους Σοσιαλιστές Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά για τις ε, συνεχείς σας προσπάθειες ε, σχετικές με την ΕΦΡΑΓ. Θα μπορούσαμε να δούμε το θέμα αυτό και κατά τη διάρκεια της εξέτασης του προπολογισμού του 2017 γιατί τα θέματα αυτά συνδέονται στενά. Υπενθυμίσατε ορθά ότι όταν υιοθετήσαμε το, τα προηγούμενα κείμενα είχαμε αναφέρει ότι θέλουμε μέσω του προπολογισμού να διατηρήσουμε μια εποπτική ικανότητα επί της εξέλιξης των δραστηριοτήτων της ΕΦΡΑΚ. Και με το ίδιο πνεύμα, προς την ίδια κατεύθυνση, θα πρέπει να συνεχίσουμε να χειριζόμαστε το θέμα του προπολογισμού της ΕΦΡΑΓ. η Επιτροπή μας θα πρέπει να παρέμβει στην ε, θέση ισχύ του πρωτύπου Ιαθαρές 9. Ε, το μήνυμα είναι ότι ετησίως ε, θα πρέπει να αξιολογούμε την κατάσταση προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει δυνατότητες παρέμβασης και να υποφελούμαστε της ψήφισης του προπολογισμού όχι για να παρέμβουμε στην ίδια την διαχείριση, την οικονομική διαχείριση, αλλά για να θέσουμε τους όρους της μεταρρύθμισης της ΕΦΡΑΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ECR. Κύριος Καμάλντα, δεν βλέπω κανέναν τον αντικαθιστά για τους ε, φιλελευθέρους. Ευχαριστώ, θα είμαι συντομότατη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Στόλογεν για την εξαιρετική έκθεση, αλλά μας έχει συνηθίσει σε εξαιρετική ε, δουλειά με τις εκθέσεις. Μας είπατε για το αντικείμενο της έκθεσης. Ε, λίγες σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, κατάλαβα καλά ότι δεν έγιναν αλλαγές από την Κομισιόν ε, σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τα ποσά που διατίθενται στην ΕΦΡΑΓ, γιατί δεν το βρίσκω στην έκθεση. Δεύτερη ερώτηση. Επαιδείο δραστηριότητας της ΕΦΡΑΓ, η Περβάνς Περές, επίσης μίλησε για την έκθεση Μάιλστατ αλλά στο ψήφισμα για το IFRS τον Ιούνιο, στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, έχουμε δώσει στην ΕΦΡΑΓ διαφορετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες κάπως εκτός ε, έκθεσης μάλιστα και είναι σημαντικό η ΕΦΡΑΓ να μπορεί να ε, ανταποκριθεί σε αυτά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αποτελεσματικά. Θα ήθελα λοιπόν να καταρτήσω μια τροπολογία που θα λέει ότι η ΕΦΡΑΓ θα πρέπει να είναι βέβαιο ότι θα παρακολουθεί και αυτά τα καθήκοντα. Όπως είπε η Φερβάνς, πρέπει να μπορούμε να αξιολογήσουμε το σύνολο του έργου της ΕΦΡΑΓ και τα καινούργια που προσθέθηκαν ε, πέρα από την έκθεση Μάιστατ. Ε, αυτό το μικρό, ε, αυτή τη μικρή προσθήκη θα κάνω στην κατά τα άλλα εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Μιγγέλ Διέγκας για την Γκουε. Ε, συμφωνούμε με την ανάγκη αύξηση της βελτίωσης ποιότητας της πληροφορίας ε, και ε, την ανάγκη για την ομογενοποίηση της πληροφορίας έτσι ώστε το σύστημα να γίνει πιο διαφανές, πιο ευανάγνωστο σε ένα κόσμο που οι οικονομικές, οι χρηματοοικονομικές πτυχές επικρατούν της πραγματικής οικονομίας. Είναι σημαντικό το σύστημα αυτό να γίνει πιο διαφανές ε, προς ε, όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά το μοντέλο διακυβέρνησης της ΕΦΡΑΚ. Το δημόσιο συμφέρον δεν εκπροσωπείται επαρκώς ε, στην ΕΦΡΑΚ ε, δεν υπάρχει μια ισοτιμία ανάμεσα στους ε, ιδιωτικούς φορείς, ε, τους ασφαλιστές, τις τράπεζες κλπ. αφενός και του κρατικού το, τομέα αφετέρου. Ούτε καν σε επίπεδο χρηματοδότησης, το 60% της χρηματοδότησης είναι κρατικό, δημόσιο. Απ' την άλλη μεριά οι κρατικοί φορείς, τα κράτη, οι κυβερνήσεις κλπ. δεν εκπροσωπούνται επαρκώς και ισότιμα έχουν ε, ούτε καν 50% των ε, θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ε, θα θέλαμε η, πράγματι έφραγ να γίνει μεσοπρόθεσμα ε, κρατικός, δημόσιος φορέας όλες οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί ε, ε που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προπολογισμό, όπως η FRES και άλλες θα πρέπει να δούμε ποιες σχέσεις έχουν μεταξύ τους και να αντιμετωπίσουμε το ίδιο ακριβώ πρόβλημα. Ε, η, το Ίδρυμα Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για παράδειγμα, ε, χρηματοδοτείται από, χρηματοδοτείται από τη Lehman Brothers. Ε, προφανώς εκεί πώ θα εκπροσωπηθεί το δημόσιο συμφέρον επαρκώ. Πρέπει, όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν παρόμοια προβλήματα. Συμφωνούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η πληροφόρηση, το σύστημα να είναι πιο ευανάγνωστο, ε, πιο διαφανέ. 3 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν. Παρ' όλα αυτά έχουμε μια αμφιβολία σε ό,τι αφορά την επαρκή αντιπροσώπευση των κρατικών συμφερόντων, των δημοσίων συμφερόντων. Ευχαριστώ. Ήρθε ο συνάδελφος Καβάλη. Ο και ο συνάδελφος Καμάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και συμπαθάτε με αλλά είχα ποντάρει στο ότι θα τα πούμε αργότερα, οπότε και άργησα και εγώ να έρθω. Ναι, δεν άκουσα αυτά που είπαν κάποιοι από τους συναδέλφους, αλλά ό,τι άκουσα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Ε, τέλος πάντων, θα τα πούμε διμερώς μετά. Για ε, θυμάμαι που λέγαμε την τελευταία θητεία τι θα γίνει με την έφρα πού θα βρεθεί η και όσον αυτό Αλφα και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι πολλές από τις μεταρρυθμίσεις εκείνες ε, ε, υιοθετήθηκαν ε, ακόμα, χρειάζεται ακόμα περισσότερη διαφάνεια όπως είπαν οι συνάδελφοι από διάφορες ομάδες και επίσης θεωρούμε θετικό ότι τώρα υπάρχει καινούριο διοικητής. Σωστά αυτά που λέμε για την περίοδο εποπτείας και επίσης θεωρούμε θετικά τα περισσότερα τα οποία έχει προτείνει ο κ. Στολόγιαν ότι θα πρέπει να κάνει πιο σφαιρική ε, έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δραστηριότητες και έχουμε επίση και την έκθεση ιδίας πρωτοβουλία της ομάδας εργασίας, παραγραφή 2 και 6. Επίσης της ε, έκθεση αυτής είναι σημαντική για τις βασικές αρχές λειτουργίας της ε, ΕΦΡΑΓ όπως για το, το πώς θα δουλεύει τέλος, πώς θα λειτουργεί. Και υπάρχουν σχετικές οδηγίες, αλλά και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που θεωρείται κάτι το βαρετό, αλλά είναι πολύ σημαντικό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα τα πούμε και στην πολιτική μας ε, ομάδα, αλλά πάντως και πάλι και πάλι συγχωρήστε με γιατί δεν ήρθα εδώ να ακούσω τι είπαν οι συνέλφοι των άλλων πολιτικών ομάδων, γιατί θα πρέπει και τη δική τους γνώμη να λάβω υπόψη. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την EFTD δεν βλέπω τη Σκιώδη, την κυρία ε, Φωνστός. Βλέπω την κυρία Κάπελ. Α, ο κύριος Γκίγκολτ. Ο κύριος Γκίγκολτ θα είναι ο τελευταίος Σκιώδης, θα λάβει το λόγο. Ο κύριος Γκίγκολτ για τους πρασίνους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Στόλογεν για την έκθεση αυτή. Ε, το θέμα αυτό σχετίζεται με την ε, επιμήκη στην παράταση της χρηματοδότησης τριών οργανισμών, τριών φορέων. Ε, θέλουμε να γίνει σαφής η άποψη του Κοινοβουλίου. Ε, σε ό,τι αφορά την ΕΦΡΑΚ, Έχουμε μια, καινούργια επικεφαλή, ε, που ο, ο κ. ο πρώην συναδελφός μα έχει αναλάβει συγκεκριμένε δεσμεύσεις. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να θέσουμε όρους, πρόσθετους όρους. Έχουμε τις αιτήσεις διαδικασίες του καθορισμού του προϋπολογισμού και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να θέσουμε οποιασδήποτε όρους και προϋποθέσεις θέλουμε. Η Περμόνος Περές ε, το είπε ήδη. Σε ό,τι αφορά την PIOB, ε, οι ανησυχίες ήταν πάντα λίγες. Οπότε το πολιτικό θέμα αφορά το κατά πόσον η παράταση θα δοθεί στην IFRS. Γιατί εκεί δεν έχουμε δει πραγματική πρόοδο σε αυτά που ζητήσαμε στην έκθεσή μας. Και δεν έχουμε και πολύ ε, και, ισχυρό μοχλό όπως είχαμε στην ΕΦΡΑΚ διορίζοντας τον πρόεδρο. Οπότε σωστά ότι θα, πρέπει να πούμε ότι στις αιτήσεις εκθέσεις που έτσι κι αλλιώς προβλέπονται από τον κανονισμό ε, ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να ενημερωνόμαστε για το πόσο έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις της έκθεσης Τόλογιαν. Αλλά θα πρέπει να, πάμε και λίγο πιο πέρα ακόμα, γιατί δεν έχουμε καμία εγγύηση για ορισμένες βασικές μας απαιτήσει. Ο κ. Καμάλ ε, το είπε χωρίς όρους να ε, δώσουμε παράταση χρηματοδότησης χωρίς καμία εγγύηση δεν βλέπω το λόγο πρέπει να θέσουμε και άλλους όρους όχι απλώς να τους υποχρεώσουμε να μας ε, αναφέρουν την πρόοδό τους κάθε χρόνο θα υποβάλω τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Και αν συμφωνήσουν οι συνάδελφοι, θα δέσουμε λίγο περισσότερο την IFRS. Ε, το ε, συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο της IFRS ε, δεν του σωστά γιατί πολλά μέλη του δεν συμφωνούν με το ρόλο τους. Και ο πρόσωπος της Κομισιόν εκεί, στο Συμβούλιο Παρακολούθησης, βρίσκεται σε μια ομάδα η οποία πραγματικά δεν θέλει να ελέγξει την οργάνωση αυτή. Και ο Μισελ Μπαγνιέ είχε υποφέρει πολύ καιρό από αυτό το πρόβλημα. Ε, ε αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα της ηγεσία ε, ε, θα δημιουργηθούν πνευματικά προβλήματα δημοκρατικής λειτουργίας. Ευχαριστώ. Κύριε Γκίγκολτ, ο εισηγητής. Ο εισηγητής ο κύριος Στόλογιαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν για την έκθεση αυτή και όλοι είναι μέλη της μόνιμης ομάδας που εστιάζει στα θέματα αυτά προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς. Ε, τώρα, λίγα πράγματα θα πω. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αποκριθεί σε κάποιες ανησυχίες μας, δηλαδή για παράδειγμα προσπάθησαν να μας δώσουν να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι το δημόσιο αγαθό για να κρίνουμε τα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Είναι σημαντικό, γιατί αν ζητήσουμε από την ΕΦΡΑΚ να λάβει υπόψη της ε, πώς θα εφαρμοστεί ένα κριτήριο, πρέπει να έχουμε και στο δικό μας το μυαλό πώς πρέπει να εφαρμόζεται το συγκεκριμένο κριτήριο. Βέβαια, δεν νομίζω ότι η δουλειά που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να συζητήσουμε την ιδέα που ε, γραπτός κατέθεσε η Κομισιόν για το τι σημαίνει δημόσιο αγαθό, για παράδειγμα, σε σχέση με κριτήρια ε, έγκρισης ε, ε, κάποιου προτύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έδωσα αυτό το παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι εκτιμώ το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάποιες ανησυχίες μας ακόμα και αν οι αντιδράσεις της δεν είναι τελεσίδικες. Ε, θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο τις ε, προτάσεις για την έφραγ. Ε, μπορούμε να επηρεάσουμε την έφραγ αφού δίνουμε τα περισσότερα κονδύλια που χρειάζεται. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε σε όλους είναι ότι στην έφραγ Ε, εργάζονται υψηλής ειδίκευσης ε, εμπειρογνώμονες και οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται σαφή εικόνα σε σχέση με τις προοπτικές χρηματοδότησης της ΕΦΡΑΓ. Γι' αυτό η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή αφού τους δίνει μια ιδέα για τα επόμενα τρία χρόνια όμως. Όπως οι συνάδελφοι έχουμε τον ετήσιο προϋπολογισμό που είναι ένα μέσον που μπορεί να βάλει stop αν η ΕΦΡΑΓ δεν συνεχίσει να εφαρμόζει όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι συστάσεις που έχουμε ενσωματώσει στο ψήφισμα το φετινό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν αφορά μόνο την ΕΦΡΑΓ αλλά και το Ίδρυμα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και ο κύριος Γκίγκολτ είπε πολλά για το Ίδρυμα αυτό. Βέβαια δεν είμαστε ευτυχείς με τις απαντήσεις του Ιδρύματος στις ανησυχίες μας. Τώρα, για το χρηματικό ποσό μιλάμε για 13,8 εκατομμύρια ευρώ που έχει μπει στην πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα αυτό. Όπως αποφασίσαμε τότε, εγκρίναμε μόνο τη χρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2016. Ο κύριος Κόρζερ, που είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΦΡΑΓ, είναι ανοιχτός σε συναντήσεις μαζί μας για να συζητήσουμε όλες τις ανησυχίες μας για τη δραστηριότητα της ΕΦΡΑ και την περαιτέρω εφαρμογή των ε, συστάσεών μας. Και ελπίζω ότι θα τιμήσει αυτή τη δέσμευση. Πρέπει να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει τώρα πολύ περισσότερο σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τα θέματα του Ιδρύματος ε, και το, τα διεθνή πρότυπα που είναι σημαντικά για την υγεία των ε, κεφαλαίων των επενδυτών και άλλων εμπλεκομένων. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευτυχής για την συνεισφορά των συναδέλφων, περιμένω τις τροπολογίες τους και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια καλή συμφωνία για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με την έκθεση αυτή. Και βέβαια θα πρέπει να αρχίσουμε και τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κιόδης Τώρα είδα ότι είναι εδώ ο πρώην συνάδελφος και έχουμε και χρόνο. Ευχαριστούμε που μας επισκεφθήκατε σήμερα. Ε, έχετε κάποιο σχόλιο να μας κάνετε μετά από αυτά που ακούσατε. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το μόνο σχόλιο είναι ότι είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι μαζί σας ξανά εδώ σε αυτήν την αίθουσα και, με, και μπορώ να υπηρετήσω τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με άλλο τρόπο και από άλλη θέση. Θα τηρήσω το λόγο μου. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλό βράδυ. 6 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Ε, καλό σας βράδυ.